Please, uh, can you be seated? Παρακαλώ καθίστε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Υπήρχε μια συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών για ένα πολύ σημαντικό θέμα και ο πρόεδρος αποφάσισε να παρατείνει κατά λίγο τη διάρκεια της. Να ξεκινήσουμε λοιπόν όσο το δυνατόν πιο σύντομα ώστε να έχουμε και αρκετό χρόνο για αυτή την πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. κύριε ε, ε, Πρόεδρε, δεν σας αφορά, όμως... Ε, ε εδώ βλέπουμε ότι όταν έξω από την πόρτα ε, περιμένουν 100 άτομα ε, για να ξεκινήσει μια συνεδρίαση ε, δεν είναι σύντημα μονάχα ευγένεια αλλά είναι και σωστή λειτουργία και από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρο μα δεν μπορεί να συγκρατήσει το χρονοδιάγραμμα και αυτή τη στιγμή έχει φύγει οπότε πρέπει να το πω σε εσά για να το μεταφέρετε. Θα περιμέναμε λοιπόν μελλοντικά να τηρεί το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν. Αυτό ακριβώς έκανα πριν από λίγο. Δυστυχώς ε, δεν διορθώθηκε το θέμα, αλλά ε, να το επαναλάβω και πάλι, διότι πραγματικά υπήρχε πολλοί κόσμος που περίμενε και πραγματικά λυπάμαι γι' αυτό. Να προσπαθήσουμε όμως να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με την ημερήσια διάταξη και το χρονοδιάγραμμα διότι όλα τα θέματα που συζητούμε είναι πάρα πολύ σημαντικά και συμφωνώ και με τον κύριο Λάγκεν ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε. Να ξεκινήσω λοιπόν καταρχάς ε, καλωσορίζοντας ε, θερμά τους ε, προσκεκλημένους μας για τη δημόσια ακρόαση για το θέμα ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην Ευρώπη και για όσους είστε εδώ και για όσους θα ακολουθήσουν αργότερα να ενημερώσω ότι η ε, συνεδρία συμμεταδίδεται ζωντανά μέσω web streaming και οπότε μένους πρέπει να τη δείτε και αργότερα. Ε, είναι ένα από τα θέματα ε, τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ στο οικονομικό θεματολόγιο, διότι αυτή τη στιγμή καλείται προσωρινό το καθεστώς του ΦΠΑ στην Ευρώπη, ε, το οποίο είναι περίεργο και από την άλλη ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σημαντικές απώλειες, οι οποίες ανέρχονται σε 150 δις ευρώ και ο Επίτροπος είναι πεπισμένος ότι η πρόταση αυτή θα μπορέσει να μειώσει ουσιαστικά αυτές τις απώλειες. Ακόμα δεν υπάρχει μια οριστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωρίζουμε όμως τι έχει τεθεί επιτάπητος και ε, στόχος αυτής της ακρόασης είναι να ακούσουμε πληροφορίες από διάφορους ενδιαφερομένους και εμπειρογνώμονες για τον αντίκτυπο και τις πρακτικές συνέπειες των προτινόμενων αλλαγών και είμαι βέβαιος ότι οι ευρωβουλευτές ε, θα υπησέλθουν και σε λεπτομέρειες. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω από κάθε πυρογνώμονα που είναι εδώ να τηρήσει το χρόνο των 5 λεπτών για την παρέμβασή του. Ε, θα περάσουμε στους κοιόδης τους για τα θέματα αυτά. Θα υπάρχουν ερωτήσεις ε, διάρκειας 2 λεπτών και μετά θα υπάρχουν δυνατότητα απαντήσεων 3 λεπτών και μετά θα έχουμε και μια διαδικασία ε, να προσπαθήσουμε λοιπόν να ε, έχουμε όσο δυνατόν περισσότερε παρεμβάσει. Δεν θέλω να σπαταλήσω άλλο από το χρόνο σα να δώσω απευθεία το λόγο στην Μαρία Έλενα Σκόπιο, η οποία είναι τιμηματάρχης ε, ΦΠΑ, Γενικός Διευθυντής Έμεση φορολόγηση και Τελωνιακή Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση. Προηγουμένω ήταν σύμβουλο του Πιέρ Σκοβισή και ταυτόχρονα έχει σπουδάσει και νομικά και ταξιδεύει ανά την Ευρώπη για να εξηγήσει τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Την ευχαριστούμε πάρα ε, πολύ ε, γιατί ήρθε και στην Πράγα και έγινε μια πολύ σημαντική συζήτηση. Ε, παρακαλώ, φροντίστε να τηρήσετε το χρόνο των πέντε λεπτών για να έχουμε και αρκετό χρόνο για συζήτηση στη συνέχεια. Ευχαριστώ και καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για μας να είμαστε εδώ σήμερα και να συμμετέχουμε σε αυτή την ακρόαση. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ για να εξηγήσω όχι μόνο το οριστικό καθεστώς, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο Πρόεδρος, αλλά και τις άλλες προτάσεις οι οποίες αποτελούν τμήμα αυτής της στρατηγικής για να έχουμε έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ. Γνωρίζετε όλοι ότι προσπαθούμε η Ευρώπη σε θέματα ΦΠΑ να έχει απλότητα, να έχει και ένα επικαιροποιημένο σύστημα για τον 21ο αιώνα θα πρέπει ε, να παρακολουθούμε όχι μόνο τις αλλαγές στην κοινωνία μας, αλλά και τις ανάγκες οι οποίες μας οδηγούν να προσπαθούμε να φροντίσουμε καλύτερα τους πόρους μας, ώστε να μην πιέσουμε πάρα πολύ σε θέματα φορολογίας, αλλά να μπορούμε να ε, ε αντιμετωπίσουμε ε, την φοροδιαφυγή και να πάρουμε ό,τι μπορούμε να αποκομίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά προτάσεις, οι οποίες αξίζει να τι αναφέρουμε. Κάποιες έχουν ήδη εγκριθεί και μάλιστα πολύ γρήγορα. Κάποιες είναι στη διαδικασία συζήτησης και κάποιε κάποιες ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί. Θα ξεκινήσω με την πρόταση ορόσημο αυτή η οποία ουσιαστικά θα δώσει τον τόνο και για όλα τα υπόλοιπα και θα συντονίσει όλες τις δραστηριότητες μας και συντόνισε και τις δραστηριότητες μας. Είχαμε πολύ μεγάλο διάσκημα μεταβατικού καθεστώτος και θέλαμε να το έχουμε αυτό το μεταβατικό καθεστώς μέχρι να υπάρχει ένα οριστικό καθεστώς το οποίο θα βασίζεται στην προέλευση αλλά αυτό που δείχνει αδύνατον. Ελήφθη λοιπόν η απόφαση να περάσουμε σε ένα οριστικό καθεστώς ε, βάσει προορισμού. Αυτό δεν είχε τεθεί σε καμία νομοθετική πράξη, ούτε καν σαν μέτρο το οποίο δηλώθηκε και αυτό εγκρίθηκε πέρσι τον Οκτώβριο και πλέον συζητάται στο Συμβούλιο. Είναι τμήμα του νέου άρθρου 402 που λέει ότι το οριστικό καθεστώς θα βασίζεται στη χώρα προορισμού και θα λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και θα έχει διακριτά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορέσουμε να συζητήσουμε φυσικά στη διάρκεια των ερωτήσεων. Πέραν αυτού προσπαθούμε τώρα το παρόν μεταβατικό κοθεστό να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Γι' αυτό είχαμε και κάποιες ε, ε, γρήγορε αλλαγέ οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και συζητιόνται τώρα στο Συμβούλιο και έχουμε και ε, την έννοια του πιστοποιημένου υποκείμενου στο φόρο. Certified Taxable Person. Είναι ένα νέο όρο στο σύστημα το οποίο θα μα επιτρέψει να έχουμε μια βαθμιδόν εισαγωγή και αυτό θα είναι μια επανάσταση τύπου Κοπέρνικου στην εφαρμογή του ΦΠΑ. Και να σας πω ότι δεν είναι μόνο μια επανάσταση τύπου Κοπέρνικου, αλλά είναι και μια φορολογική αναγέννηση, διότι μαζί με αυτό είχαμε και μια σειρά από άλλες προτάσεις, οι οποίες συμπληρώνουν αυτή τη βασική αλλαγή. Άλλες προτάσεις, οι οποίες στόχο έχουν να κάνουν το σύστημα Πλούστερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, που εγκρίθηκε και τον Ιανουάριο φέτος η σχετική πρόταση και κάποια ε, συνοδευτικά μέτρα για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η στάθμιση και αυτό ε, εγκρίθηκε και επίσης τον Ιανουάριο. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δέσμης μέτρων όμως είναι τα νέα μέτρα για τη διοικητική συνεργασία. Αρχές και πολιτικές που είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται είναι πολύ πιο σημαντικός. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε στις χώρες μας τα εργαλεία και τις δυνατότητες να συνεργάζονται αποτελεσματικά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ε, το μοντέλο που προσπαθούμε να σχεδιάσουμε θα εφαρμόζεται εφαρμόζεται ε, με επιδεξιότητα στην πράξη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μόλις εγκρίθηκε από την Επιτροπή το Δεκέμβριο και τώρα συζητιέται με πολύ επικοδομητικό πνεύμα ε, στο Συμβούλιο. Ε, προσβλέπουμε σε ταχεία έγκριση και αυτό γίνεται προς το συμφέρον των κρατών μελών, προς το συμφέρον των πολιτών που καταβάλουν τους φόρους τους και προς το συμφέρον των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που αποτελούν τμήμα της κοινωνίας μας, της οικονομίας μας. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά τα διάφορα μέτρα θα πρέπει να θεωρηθούν ως σύνολο, να θεωρηθούν ως μια κοινή προσπάθεια προς ε, τη διαμόρφωση ενός εντελώς καινούριου συστήματος ε, ΦΠΑ. Και να σας πω και τα καλά νέα εγκρίθηκε μετά από πολύ καιρό ομόφωνα το σύστημα νέων κανόνων για το πώ θα εφαρμόζεται ΦΠΑ για τι εξαποστάσεω πωλήσει, που είναι ε, η επέκταση τη αρχή που θέλουμε να εφαρμόσουμε και για το οριστικό καθεστώ, το οποίο αποκαλείται ε, μόνο απευθυντική φυρίδα One Stop Shop. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω σε ερωτήσεις. Thank Ευχαριστούμε εμείς για την ενημέρωση και γιατί τηρήσατε και το χρόνο αγόρευσης. Επόμενη ομιλήτρια. Έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε την Ρίτα Ντελαφέρια, καθηγήτρια και η Δήμονα περί τα φορολογικά, το λέω εγώ, αλλά το λέει και το International Tax, Tax Review πριν δύο χρόνια την ε, κατέταξε στους ε, ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στα φορολογικά ζητήματα. Η κυρία Τελαφέρια είναι καθηγήτρια φορολογικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Leeds και International Research Fellow στην Οξφόρδη και στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνα στη χώρα της ε, σκέπτρια ε, καθηγήτρια. Έχετε έρθει σε ακροάσεις εδώ και όταν ε, ήμασταν στο Λονδίνο επίσης σας ακούσαμε σε μια ακρόαση εκεί. Θα σας ξανακούσουμε σήμερα, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Τελαφέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να σχολιάσω τις ε, προτάσεις. Το βασικό ε, θέμα της σύντομης αυτής παρουσίασης, η εισαγωγή, αν θέλετε, είναι οι συντελεστές ΦΠΑ, το συγκεκριμένο στοιχείο της πρότασης. Πριν περάσω όμως στους συντελεστές, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαδικασία σχετικά με τη θέσπιση ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ το διδακτορικό μου λεγόταν ακριβώς Reckon with Transition, πώς δηλαδή θα πετύχουμε τη μετάβαση. 30 χρόνια μας χρειάστηκε, αλλά φαίνεται ότι πλέον τα καταφέραμε και ε, ελπίζω στους επόμενους μήνες και όχι χρόνια να επιτύχει η προσπάθεια της Κομισιόν. Αυτό που με ανησυχεί πολύ περισσότερο είναι η πρόταση για τους συντελεστές ΦΠΑ. Δεν θα επισέλθω στις ε, ε, μεγάλες λεπτομέρειες και το ιστορικό του συστήματος ΦΠΑ. Ούτε και θα ήθελα να μακρηγορήσω για τις νομικές και οικονομικές συνέπειες ε, των συντελεστών ΦΠΑ. Βέβαια, έχω διαβάσει στην Επιτροπή σας ε, μερικά άρθρα που έχω συγγράψει για το θέμα αυτό, ελπίζοντας να είναι ένα υπόβαθρο και για τη σημερινή συζήτηση. Ο πρωταρχικός μου σήμερα στόχος είναι να σας δώσω το πλαίσιο για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το που βρισκόμαστε σήμερα και να προειδοποιήσω για τους σημαντικούς κινδύνους που κατά την άποψή μου ενέχει η πρόταση. Προσπαθούμε να αναρμονίσουμε το σύστημα ΦΠΑ και τους συντελεστές ΦΠΑ εδώ και 50 χρόνια από τη δεκαετία του 60, 1960. Έρχονται και, έρχονται και νέες προτάσεις συνεχώς και συνεχώς προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μία δομή για το ΦΠΑ. Η πρόταση η τωρινή της Κομισιόν συνιστά ε, μία ρηξικέλευτη αλλαγή. Αν εγκριθεί αυτή η πρόταση θα οδηγήσει σε κατάργηση της αναρμονισμένης προσέγγισης. Το, το επιχείρημα που προβάλλει η Κομισιόν για την αλλαγή αυτή θέσης και στάσης είναι ότι το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ δεν απαιτεί την εναρμόνιση των συντελεστών ΦΠΑ. Εγώ διαφωνώ κάθετα και με την αρχή αλλά και με το συμπέρασμα επομένω. Η αρχή, το αξίωμα είναι ότι με το οριστικό καθεστώ ΦΠΑ δεν έχουμε πλέον διασυνοριακέ αγορέ, δεν χρειάζεται κατά συνέπεια και εναρμόνιση. Είναι γεγονό ότι με το οριστικό αυτό σύστημα θα σταματήσει ε, η διασυνοριακή πόλη στο το cross-border shopping. Αυτό δεν σημαίνει όμως πρέπει να σταματήσει και η εναρμόνιση. Όπως αναγνωρίζει η Κομισιόν, αν εγκριθεί αυτή η πρόταση, θα δώσει την ελευθερία στα κράτη-μέλη να μπορούν να αλλάζουν τους συντελεστές τους. Κάτι που αναπόφευκτα και κατά ανάγκη θα αυξήσει τις διαφορές στους συντελεστές ΦΠΑ ανά την Ευρώπη. Επίσης, κατά την άποψή μου, επίσης αναπόφευκτα, θα οδηγεί σε διάβρωση της βάσης που σημαίνει κάποια στοιχεία θα βγαίνουν από το κανονικό ΦΠΑ και θα έχουμε μειωμένους συντελεστές. Οι πολιτικο-οικονομικές επιπτώσεις ε, μιας τέτοιας μετακίνησης είναι προφανής για εμάς που εργαζόμαστε στον κλάδο. Επί σειρά ετών τα κράτη-μέλη πιέζουν για αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ και παρότι δεν το γνωρίζω με τα βεβαιότητα, υποπτεύομαι ότι αυτό έχει ε, μεταξύ άλλων κινητοποίηση και την Κομισιό για να καταθέσει αυτή την πρόταση. Όμως η οικονομική πίεση που τώρα ε, ασκείται θα είναι πολύ εντονότερη στη συνέχεια. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούν να πούν είναι μπορούμε να το αλλάξουμε λόγω των κανόνων της Ένωσης. Από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει αυτή η αναμόνηση, δεν θα μπορούν να κατηγορούν τους κανόνες της Ένωσης και η πολιτική πίεση για αφαίρεση κάποιων στοιχείων από τη βάση δεν θα είναι εύκολο κανείς να την παραγνωρίσει. Η χρήση μειωμένων συντελεστών και διάβρωση της βάσης ε, μπορεί κάποιοι να πούν ότι είναι καλή πολιτική, αλλά δεν είναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ο λόγος για τον οποίο εφαρμόζονταν οι συντελεστές αυτοί ήταν ουσιαστικά δύο, είτε μαζί είτε ένας εκ των δύο, για την προστασία των φτωχότερων οικοκυριών και συμπολιτών μας και ο δεύτερος λόγος ήταν η αύξηση της χρήσης ειδών ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Κάθε φορά που προσπαθούμε εμπειρικά να μετρήσουμε τις μειώσεις στις τιμές, συνέπεια της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ δεν βγάζουμε αποτέλεσμα. Είναι πολύ μεγάλη αντίσταση της αγοράς και τι γίνεται τελικά. Οι λιανοπολιτές απορροφούν τις ε, μειώσεις αυτές. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στην πράξη είναι ότι επιδοτούνται συγκεκριμένοι τομείς. Επίσης, αλλά και να δούλευε το σύστημα και να μειώνονταν οι τιμές, θα είχαμε μια άλλη συνέπεια. Αν δούμε τα μοντέβα κατανάλωσης και για τα βασικά είδη, οι πλουσιότεροι συμπολίτε μας είναι αυτοί που καταναλώνουν περισσότερο. Ψωμί, γάλα, οι πλούσιοι καταναλώνουν περισσότερα από αυτά τα προϊόντα. Τι συμβαίνει λοιπόν ουσιαστικά, μειώνουμε την, ε, τους φιόλου για τους πιο πλούσιους. Από στατιστικής πλευράς ε, ε, μπορεί αυτό να μην έχει νόημα, αλλά οι πλουσιότεροι είναι αυτοί οι οποίοι ωφελούνται από τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ ανεξαρτήτως ε, ε, του είδους αυτού. Μπορεί να είναι φρούτα, μπορεί να είναι ψώμα, μπορεί να είναι γάλα. Οι πιο πλούσιοι θα ωφεληθούν και θα υπάρξει απόλυση οδήματο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των φτωχότερων συμπολιτών μέσω των συστημάτων κοινωνική προστασία. Για όλου αυτού του λόγου, η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ μπορεί να φαίνεται ελκυστική, αλλά δεν είναι πανάκια, που είναι και στόχος. Και το τελευταίο, που έχω να πω είναι ότι παρά το, μάλλον πέραν των οικονομικών και νομικών συμβαίνει και κατά την άποψή μου αντισυνταγματική αυτή η πρόταση, διότι δεν θεωρώ ότι μπορεί να ενταχθεί στην νομική βάση που είναι το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαιτεί η νομοθεσία που εγκρίνεται για στόχους ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ε, ως στόχο την εναρμόνιση και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, κάτι που δεν επιτυγχάνει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο σκέλος, κατά την άποψή μου, επιτυγχάνεται. Και ολοκληρώνω με μια φράση που αρέσκομαι να χρησιμοποιώ σε τέτοιου είδου ε, εισαγωγικέ ομιλίες μου. Το 1985 Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν πρότεινε λευκή βίβλο για θέσπιση τη ε, ε, Οικονομικής Ένωση, είπε ότι η κοινότητα τώρα θα πρέπει να κάνει ένα ακόμη βήμα να κάνει κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να προδώσει την εμπιστοσύνη να ακολουθεί στα, τις επιταγές των ιδρυτών της Ένωσης, των πατέρων της Ένωσης και να μην οδηγήσει σε ένα λιγότερο ευημερές μέλλον από αυτό το οποίο θα ε, είχαν αλλιώ. Και θα πρέπει να έρθουμε στο ύψος της πρόκλησης. Το 1985 αυτό είχε ε, ήταν απόλυτα σωστό, εξίσου σωστό είναι και σήμερα. Ξέρω ότι πάει ίσως ενάντια στη λογική σας αυτό που σας λέω και ζητώ να κάνουμε ένα άλμα ε, πίστης, ε, αλλά πρέπει να αρθούμε στο ύψος των προκλήσεων και να έχουμε βάσεις γερές οικονομικές και νομικές για να κάνουμε προτάσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Μεγάλη ήταν η πρόκληση στα λόγια σας. Παρακολουθούσα με μεγάλη προσοχή και έχασα το χρονόμετρο, αλλά... Εκτός σχολείου, ε, εκτός του σχολείου, τέλος πάντων δυστυχώς αρχίσαμε 25 χρόνια αργότερα. Επόμενη είναι η Λεζέ. Πάνω από 30 χρόνια ασχολείται από το Law Square, συνάδελφος με τα φορολογικά ζητήματα και για τη επίλυση διαφορών φορολογικών. Τώρα περνάμε λοιπόν στη δικηγορική σκοπιά, αφού ακούσαμε την Κομισιόν και τους φοροτεχνικούς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη που με προσκαλέσατε σε αυτή την ε, συνάντηση. Ε, ζητήθηκα να μιλήσω για τους πιστοποιημένους φορολογούμενους ε, και θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια του συστήματος ε, ΦΠΑ είναι οι φοροσυλλέκτες οι οποίοι δεν αμείβονται και έχουμε 357.000 τέτοιους φοροσυλλέκτες ε, πολλοί εξ αυτών ασχολούνται με το ε, διασυνοριακό εμπόριο και το 50% εξ αυτών ε, γίνεται μεταξύ ομάδων επιχειρήσεων λόγω των ολοκληρωμένων αλυσίδων παροχής και θα πρέπει λοιπόν να εισάγουμε δύο κατηγορίες μη αμοιβόμενων φοροεισπρακτών και μόνο οι πιστοποιημένοι ε, θα μπορούν να υποφεληθούν από την συγκεκριμένη απλοποίηση την απόδειξη της εξαίρεσης ε, για παράδειγμα και στο πρώτο στάδιο του τελικού καθεστώτος θα μπορούν να αγοράζουν ε, διευρωπαϊκά αγαθά χωρίς επιπλέον χρέωση. Η απάντησή μου σε αυτό είναι όχι. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω ορισμένους λόγους και μερικούς από αυτούς τους συμπεριέλαβα και στο έγγραφο το οποίο κατέθεσα κάποιες ανησυχίες. Αν είσαι ε, ε, πιστοποιημένος, ε, εγκεκριμένος οικονομικός ε, ε, παράγοντας, τότε υπάρχουν κάποιοι όροι οι οποίοι πρέπει να ακολουθηθούν και οι οποίοι απέχουν από την πρόταση που κατατέθηκε. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό. Δεύτερον, θα περιλαμβάνει ένα ε, κόστος ε, στο νόμιμο έμπορο και μπορεί να δημιουργήσει φραγμούς και ε, περιορισμούς ε, στο εμπόριο και στην επιχειρηματικότητα ιδιαίτερως για τις start-up, τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης κάθε φορά που κάνω μια συναλλαγή δεν χρειάζεται μονάχα να επιβεβαιώσω εάν ο πελάτης μου είναι ικανοποιημένος από το ΦΠΑ, καλυμμένος από το ΦΠΑ αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσω και αν ε, ο πελάτης μου έχει το στάτους ε, του πιστοποιημένου φορολογούμενου. Ε, χρειάζεται λοιπόν αυτό για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή. Και τέλος υπάρχει ένας κίνδυνος διότι η παροχή τέτοιου στάτους θα, σε περίπτωση που οι κανόνες δεν εφαρμόζονται υπό ίδιους κανόνες θα δημιουργήσει ένα νέο ε, πλαίσιο όταν επιλέγουμε την τοποθεσία ε, της επιχείρησης. Δηλαδή θα έχουμε CTP ε, shopping ε, και επίσης μπορεί να έχουμε περιπτώσεις όπου ε, απαταιώνες μπορεί να είναι ιδιαίτερα καινοτόμοι χρησιμοποιώντας αυτό το ε, πιστοποιητικό εις του συστήματος ΦΠΑ και του εμπορίου και στη συνέχεια άλλο θέμα το οποίο έχουμε είναι ότι εισάγουμε ε, τουλάχιστον στο, ε, στο τελικό σύστημα διασυνοριακό ΦΠΑ θα συλλέγουμε είτε το ΦΠΑ είτε αν υπάρχει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ως καταναλωτής ε, και στο άλλο σενάριο ε, θα πρέπει ε, να έχουμε την αρχική χρέωση και έτσι λοιπόν έχουμε εξαιτία αυτού του διπλού στάτους τον κίνδυνο να δημιουργούνται προβλήματα. Οπότε ποια είναι η εναλλακτική. να επιλύσουμε τα ε, βασικά αίτια της απάτης ε, ΦΠΑ. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το μοντέλο ε, καταγραφής των επιχειρήσεων θα πρέπει ε, να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα ΦΠΑ οπότε όποτε κάποιος ε, καταγράφεται τότε θα λαμβάνει το, τη σφραγίδα ποιότητας ε, ότι είναι πιστοποιημένος φορολογούμενος και έτσι θα αποφεύγουμε τυχόν απαταιώνες Ίσως ε, να σας ακούγεται ομό, αλλά όταν έχω μία άδεια οδήγησης, για παράδειγμα, μπορώ να οδηγήσω τόσο στους εθνικούς όσο και στους διεθνείς δρόμους και αν κάνω κάτι παράνομο, λάθος, ε, τότε ή μου παίρνουν το δίπλωμα για κάποιο ε, χρονικό διάστημα ή ίσως και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έτσι λοιπόν αυτό γίνεται για να προστατευθούν οι άλλοι χρήστες, οδικοί χρήστες ε, χρειαζόμαστε λοιπόν στο χρονικό διάστημα που έχουμε από τώρα έως το 2022 ε, να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο ε, ευρωπαϊκής καταγραφής και ε, κάνοντας αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να αξιολογούμε το πώς μπορεί ε, να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ε, της, της καταγραφής των πιστοποιημένων φορολογουμένων. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι εισέρχονται ενώ αυτοί οι οποίοι είναι ήδη στο σύστημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία που ήδη υπάρχει. Ας κάνουμε όλο αυτό, ας μοιραστούμε ε, τη ικανότητα αυτών των πιστοποιημένων φορολογουμένων, να μοιραστούμε τα δεδομένα από ε, αυτούς και φυσικά χρειάζονται και κυρώσει. Αν κάποιο κάνει κάτι παράνομο, ε, μπορεί να συσχετιστεί αυτό με την οδηγία PIF. Εάν έχουμε σοβαρές παραβάσεις, τότε μπορεί να άρεται η πιστοποίηση, μπορούμε να ε, πάβουμε την ε, καταγραφή και έτσι λοιπόν θα έχουμε ε, μία βάση δεδομένων νόμιμων εμπόρων. Και φυσικά χρειαζόμαστε μία περίοδο μετάβασης, θα έχουμε χρόνο να το φροντίσουμε αυτό. Κλείνοντας λοιπόν, χρειαζόμαστε άμεσες επιδιορθώσεις, όμως όχι με τους πιστοποιημένους φορολογούμενους, χρειαζόμαστε ε, το ολοκληρωμένο καθεστώς ε, και ας αρχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε έναν μηχανισμό που καταγραφεί ταυτότητας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μέσω ενός νέου συστήματος για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε, να προστατεύσουμε τους νόμιμους εμπόρους απέναντι στους απαταιώνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Κριστιαν Κοτ ο οποίος είναι πρόεδρος του Business Europe του Τμήματος Πολιτικής ΦΠΑ και ασχολείται με θέματα ΦΠΑ εδώ και 15 χρόνια και έχει και εκτεταμένη φορολογική εμπειρία γιατί ήταν σύμβουλος ε, φορολογικών θεμάτων στην KPMG αν δεν κάνω λάθος. Έχετε το λόγο λοιπόν και εσείς για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευγενική πρόσκληση να μιλήσουμε για το πολύ σημαντικό θέμα του μέλλοντος του ΦΠΑ. Με την Business Europe γνωρίζουμε βεβαίως πώς έχει το τρέχον σύστημα ΦΠΑ, το οποίο συστήθηκε πριν από 25 χρόνια και είναι απόλυτα κατακαιρματισμένο και αυτό σημαίνει ότι είναι ανοιχτό σε απάτη και η επιτυχία της εσωτερικής αγοράς για να μπορέσει να ε, δώσει κίνητρα για το ε, εμπόριο έχει πιέσει το τρέχον σύστημα ΦΠΑ. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο έχουμε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα δέσμες μέτρων για τη δίκαιη φορολόγηση 1, 2 και 3 είτε είναι για τους συντελεστές ΦΠΑ, το οριστικό σύστημα, τον πιστοποιημένο φορολογούμενο ή την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ είναι μια μοναδική ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ότι το νέο σύστημα θα είναι πιο απλό, θα υπάρχει λιγότερη δυνατότητα απάτη και θα προωθεί το διασυνοριακό εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σε αυτή τη συζήτηση είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε λύση να μειώνει και το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη-μέλη, καθώς επίσης και να φροντίζει και τις ε, ροές ε, μετρητών που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουμε μια γραφειοκρατία με ένα άλλο σύστημα γραφειοκρατίας. Χρειαζόμαστε όμως το οριστικό καθεστώς για να έχουμε και μειωμένη συμμόρφωση και μείωση του διοικητικού κόστους και ε, ταυτόχρονα να μειώσουμε και την απάτη. Και αυτό μπορεί να αποβεί και ιδιαίτερος περίπλοκο. Ένα βασικό στοιχείο, και όσες φορές και να το πω δεν αρκεί, ένα βασικό στοιχείο λοιπόν, οποιασδήποτε πρότασης ε, προωθήσουμε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών. Κάποιες από τις παρούσες ε, διαφορές αυτή τη στιγμή οφείλονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη της ε, φορολογικής ε, διοίκησης ενό κράτους μέλους για τη συλλογή του ΦΠΑ μας. Εάν δεν βρούμε έναν τρόπο να γεφυρεώσουμε αυτό το χάσμα, θα είναι αδύνατο να υπάρχει ένα απλούστερο σύστημα ΦΠΑ. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν αφορά μόνο την εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών, αλλά και μεταξύ φορολογικών διοικήσεων και επιχειρήσεων, νόμιμων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή. Βάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των εκτιμήσεών τη, ε, περίπου 1-3 ε, ΦΠΑ συλλέγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Αυτό ισοδυναμεί με 7% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποδεικνύει ότι ακόμα και οι πιο μικρές αλλαγές στο σύστημα ΦΠΑ μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο για την οικονομική απόδοση Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών. Το εμπόριο μεταξύ φορολογητέων επιχειρήσεων ε, υπόκειται σε ΦΠΑ και αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε σύστημα υπάρχει θα πρέπει να διευκολύνει την ομαλή διεξαγωγή αυτών των εκατομμυρίων των καθημερινών συναλλαγών και αυτή είναι η άλλη διαφορά μεταξύ ΦΠΑ και άλλων φόρων πρέπει να είμαστε σε θέση να βρούμε το κατάλληλο ποσοστό να εκδίδεται τιμολόγιο τη στιγμή της ε, συναλλαγής. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε τις συναλλαγές γιατί πρέπει να βρούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα ΦΠΑ. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος ε, ΦΠΑ, που είναι ένας ε, φόρος ο οποίος βασίζεται στις συναλλαγές. Και οτιδήποτε ε, τέτοιο έχει και κόστος για τις καθημερινές συναλλαγές μπορεί να βοηθήσει να οδηγήσει και σε σημαντικό κόστος και απασχόλησης και εισόδων. Όσον αφορά το οριστικό σύστημα ΦΠΑ, η Business Europe υποστηρίζει τη μετάβαση του συστήματο σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στον τελικό προορισμό, αλλά προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα θα πρέπει να υπάρχουν απλοποιήσει και εύκολη πρόσβαση σε ε, αξιόπιστε και σημαντικέ πληροφορίε για του κανόνε και τι διοικητικέ πρακτικέ στα άλλα κράτη-μέλη. Εάν ακολουθήσουμε τον κανόνα της χώρας προορισμού, τότε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε και να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες για το συντελεστή ΦΠΑ. Όσον αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ, υποστηρίζουμε ιδιαίτερα τι προσπάθειε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει περαιτέρω και να διευρύνει το, τη μονοπευθυντική θηρίδα που είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο ενός συστήματος που θα βασίζεται στη χώρα προορισμού και αυτό θα είναι και η πιο σημαντική απλούστευση για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει διότι η βασική πρόκληση κατά το διασυνοριακό εμπόριο είναι ε, η εγγραφή τους και, ε, και να, πώς μπορούν να αντιληφθούν τους κανόνες ΦΠΑ στο άλλο κράτος μέλος. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία όμω ε, για το στόχο τη απλούστευση των καθημερινών συναλλαγών των επιχειρήσεων και με την εισαγωγή και ενό ευρύτερου ε, συστήματο μονοαπευθυντική ηρίδα. Για παράδειγμα, ο πιστοποιημένος φορολογούμενος ε, που προτείνεται προσπαθεί να απαντήσει στην ανάγκη για απλοποίηση, αλλά η έννοια του πιστοποιημένου φορολογούμενου από μόνη τη επιβαρύνει και τι επιχειρήσει και τι φορολογικέ διοικήσει και μπορεί τελικά να έχουμε ένα πιστοποιημένο αιώνα. Ε, σε θέματα ΦΠΑ που το είπε και η συνάδελφος εκ Επιτρέψτε μου λοιπόν να επισημάνω ότι βάσει της αξιολόγησης αντικτύπου της ε, προτινόμενης ε, διοικητικής συνεργασίας το 80% της διασυνοριακής απάτης έγινε από το οργανωμένο έγκλημα και όχι από συνήθεις επιχειρήσεις. Και αυτό φυσικά είναι τελείως διαφορετικό αντικείμενο και έχουμε να παλέψουμε κάτι τελείως διαφορετικό και δεν είναι συνήθι απάτη ΦΠΑ. Τώρα για την πρόταση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, η Business Europe απογοητεύτηκε από τη φιλοδοξία τη πρόταση, γιατί στην ουσία αφορά πολύ μικρέ επιχειρήσει. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίω ότι οι πρωτοβουλίε μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να συνδέονται και με τι απλοποιήσει που προσφέρονται ε, στο πακέτο νομοθεσία B2C, ε, αλλά να υπάρχουν και απλοποιήσει ε, στι αναλυτικέ διατάξει που θα αναφέρονται στο οριστικό καθεστώ, αλλά η πρόταση δεν ε, αντιμετωπίζει πώς οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αυξηθούν στο σύστημα ΦΠΑ, εισάγοντας ουσιαστικά τις απαιτήσει συμμόρφωσης. Και ένα από τα βασικά στοιχεία το οποίο θα αναζητήσουμε είναι η αρχή και ενός ελέγχου στη χώρα έδρας. Ε, αλλά αυτό φυσικά θα επιτρέψει να γίνεται έλεγχος στο κράτος μέλος της έδρας τους ε, από άλλο κράτος μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. τελευταίο ο Γκέρχαρτ Χούμερ από την Αυστρία. Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και φυσικά επειδή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς θα επηρεάσει τις μικρές επιχειρήσεις, φορολογική συμμόρφωση ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θέλω να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποια ε, στα όσα είπε ο συνάδελφος από την Business Europe, ε, εστιάζοντας πιο πολύ στη σκοπιά των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδίω ε, δε οι μικρές επιχειρήσεις αλλά και οι ΜΜΕ έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κόστος συμμόρφωση από τις μεγάλες επιχειρήσεις Γι' αυτό υποστηρίζουμε το ειδικό καθεστώς ε, για τις μικρές επιχειρήσεις και την πρόταση για εξαιρέσεις ε, για τις νορικές δραστηριότητες την επικροτούμε πάντα για τις μικρές επιχειρήσεις ε. και ελπίζουμε ότι η απλούστευση θα ωφελήσει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ακόμη και αν δεν υπάρχει εξαίρεση. Καταλαβαίνω κάπως που οι μη πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτοί που δεν είναι εθνικές επιχειρήσεις ίσως να είναι απογοητευμένοι. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό μικρών επιχειρήσεων οι οποίες καλύπτονται από τις προτάσεις αυτές και σίγουρα υπάρχουν ε, προβλήματα ε, ανταγωνισμού αν κάποιες επιχειρήσεις ωφελούνται και κάποιες δεν ωφελούνται. Αυτό έχει να κάνει με τις τοπικές, τοπικά παρεχόμενες, παραδείγματος χάρη, υπηρεσίες, όταν έχουμε δηλαδή μεγάλο κόστος, ε, μεγάλο πλεονέκτημα, ε, ανάλογα με τα ανώτατα όρια, επειδή μπορεί να επηρεαστούν οι επιχειρήσεις με ένα πολύ ψηλό συντελεστή. Εμείς συμφωνούμε με τις 100.000 ως ε, τζίρο, αλλά σε ό,τι αφορά τις 85.000, την πρόταση για τις εθνικές δηλαδή εξαιρέσεις, ε, πολλά από τα κράτη, τα μέλη μας δεν είναι ικανοποιημένα. Καταλαβαίνουμε τη λογική. Γιατί παίρνουν ε, ένα νότατο που θα καλύπτει τα 27 κράτη-μέλη και όχι πλέον και το ΕΒ. Όμως όταν έχουμε 25.000 30.000 ευρώ ανώτατο όριο σε κάποιες χώρες και σε κάποιες επιχειρήσεις, υπάρχει φόβος, αν έχουμε 85.000 ευρώ στην νέα οδηγία, ότι θα υπάρξει τεράστια πίεση για αύξηση ανώτατου αυτού όριου και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των μελών της Ένωσής μας. Ε, ίσως λοιπόν καλό θα ήταν ε, να, έχουμε υπόψη και το εξής. Μήπως δεν χρειάζεται ανώτατο και να αφήσουμε την απόφαση να τη λαμβάνουν σε εθνικό επίπεδο τα κράτη-μέλη, αποφεύγοντα χώρε όπω το Βέλγιο ή η Γερμανία να δεχτούν πιέσει για να, ασκεί, να αυξήσουν τα σημερινά ανώτατα όρια. Και οι πιέσει να προέρχονται από τη, το, την πολιτική. Το πιο υψηλό δατόριο για τι εξαιρέσει μπορεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό, ιδίω όταν έχουμε ψηλή ένταση εργασία η ΑΠΜΕ θα συνιστούσε προσοχή με μια τέτοια διάταξη. Υπάρχει όμως μια άλλη ιδέα. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τις νοφείς επιχειρήσεις που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους, μήπως πρέπει να τις βοηθήσουμε να ενταχθούν στο σύστημα και έρχομαι εδώ στο εθνικό επίπεδο με ένα ανώτατο όριο που θα μειώνεται. Δηλαδή, μέχρι δύο χρόνια να υπάρχουν ε, περισσότερα περιθώρια εξαιρέσεων για τις έψιλων ε, Κάποιες μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές και αν θέλω να παραμείνουν έτσι, αν μην θέλουν να ψηθούν. Άρα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όρετο τα επόμενα ε, χρόνια. Να έχουμε τώρα τη μεταβατική περίοδο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνά το κατωτόριο. Θέλουμε να εξακολουθήσουν να ισχύσουν οι εξαίρεσεις για ακόμα ένα έτος. Κάποιες επιχειρήσεις όμως που είναι μέλη μας θεωρούν ότι οι τρέχουσες προτάσεις με αυτό το κατωτόριο για την πέρβαση του 50% ίσως είναι λίγο υπερβολικό. 33 ή 25% θα ήταν ένα πιο αποδεκτό όριο. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση, χαιρετούμε την θέσπιση ενός ε, κατώτατου ορίου ώστε να έχουμε ε, μέτρα απλούστευσης ε, για την καταχώρηση, την τήρηση βιβλίων, να έχουμε μικρότερες φορολογικούς περιόδους. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο τα 2 εκατομμύρια ευρώ που είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών θα έπρεπε να γίνει 5 εκατομμύρια παράδειγμα, γιατί είναι λίγο χαμηλό αυτό το ποσό. μια πρόταση για τα ευέλικτους ε, συντελεστές. Υπογράψω αυτό που άφησα από την Business Europe. Και για μας, αυτοί οι ευέλικτοι συντελεστές συνιστούν ε, μεγάλη απέτηση. Είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα της ΜΜΕ. Μόνο αν είναι εύκολο να καταλάβει οι μικρόμεσες επιχειρήσεις ποιος είναι ο συντελεστής που εφαρμόζεται σε μια άλλη χώρα και να ενημερώνεται για την αλλαγή των συντελεστών. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να μπαίνουμε σαφώς στο σύστημα για να βλέπουμε αν υπάρχουν αλλαγές. Και τελευταία πρόταση για αυτό το CTP, τον ε, υποκείμενο σε φόρο τον πιστοποιημένο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται αν είναι πολύπλοκα τα κριτήρια και πολύπλοκα τα συστήματα για το πιστοποιημένο αυτόν φορολογούμενο. Οι ΜΜΕ που μπορεί να έχουν πάει καλά κατά το παρελθόν ε, θα είναι συγκριτικά μεγάλο το μειονέκτημά τους αν δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα. Γιατί αν πληρώνει το ακόμα και αν σου επιστρέφεται, έχει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα ταμιακή ροή από τι επιχειρήσει εκείνε ε, που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ε, το σύστημα τη αντίστροφη χρέωση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλο τη ακρόαση. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο σε τέσσερι συναδέλφου μου βουλευτέ που είναι εισηγητέ και συνεχεία θα ακολουθήσουμε με τη διαδικασία Catch the Eye, προσέλκυση προσοχής του Προέδρου. Ο Φαντεν Καντελάρε από το ΕΛΚΟ εισηγητής δεν είναι εδώ. Εγώ θα τον αντικαταστήσω. Τρία ε, ζητήματα για τα οποία θέλω τα σχολιά σας. Το πρώτο μιλάμε για την φορολογική απάτη, αλλά υπάρχει και θέμα εμπιστοσύνης, έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογικών αρχών και κρατών μελών. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, στρατηγική πρωτοβουλία ίσως από κάποια κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστεί με την αντίστροφη χρέωση το πρόβλημα με τα κενά στα φορολογικά είσοδα από ΦΠΑ, ποια είναι τα ωφέλη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι από το σύστημα που την Κομισιόν. Και το τρίτο, μια ερώτηση για την Κομισιόν ξεκάθαρα, πόσο εφικτό είναι να προχωρήσει η πρόταση δεδομένου ότι χρειάζεται η συμφωνία των κρατών μελών. Και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Μήπως, δηλαδή, μήπως τραβήξει πολύ σε μάκρος η διαδικασία αυτή και δεν ολοκληρωθεί ποτέ. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Καταρχάς, ίσως η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Πόσο χρόνο έχω, παρακαλώ. Τέσσερα λεπτά. Αλλά επειδή τα πάμε καλά με τον χρόνο, εντάξει. Ίσως λίγο παραπάνω με μακρηγορήσετε. Ευχαριστώ. Γιατί θα ήθελα με την ευκαιρία να απαντήσω και σε κάποια σχόλια ε, από τους επόμενους ομιλητές από μένα. Δεν θα μακρηγορήσω. Καλό είναι πάντως να ξεκαθαρίζουμε κάποιες παρανοήσεις. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν. Για να ξεκινήσω με τους μειωμένους συντελεστές. Ποτέ δεν ενθαρρύναμε την αυξημένη χρήση αυτών των μειωμένων συντελεστών ή την ε, δυνατότητα μείωση των ε, εφαρμοζόμενων σήμερα συντελεστών. Υπάρχει αυτό ο κατάλληλο γιατί έρχε κατά κράτη-μέλη, τέλο πάντων η Κομισιόν ήθελε να προχωρήσει σε ένα οριστικό καθεστώ ΦΠΑ βάση προορισμού. Εκεί που είναι εγκαταστημένο ο προμηθευτή. Αυτό δεν θα οδηγούσε σε διασυνοριακέ πωλήσει γιατί εκεί ε, έχουμε τη μετακίνηση ενός καταναλωτή από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε στρεβλώσεις ε, στην ε, έδρα, στον τόπο εγκατάστασης. Ε, αν έχουμε την αρχή του προορισμού και διαφορετικού συντελεστέ, κάποιο μπορεί να επιλέξει τη χώρα που θα έχει χαμηλού φορολογικού συντελεστέ. Άρα, για να έχουμε δυνατόν όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφου ε, συντελεστέ, Έχουμε μια λίστα υπηρεσιών αγαθών για μειωμένου συντελεστέ. Αυτό καταρτίστηκε όταν θεσπίσαμε το προσωρινό καθεστώ ΦΠΑ. δυστυχω συναδευόταν συνοδευόταν από κάποια διακριτική μεταχείριση. Παραδείγματο χάρη, εννέα κράτη-μέλη που είχαν παρεκκλήσει, εξαιρέσει, στη δική του ε, νομοθεσία περί ΦΠΑ είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν συντελεστέ μειωμένου πέραν του καταλόγου αγαθών και υπηρεσιών που ίσχυαν για όλα τα κρατημέρια. Και εξακολουθούν να έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Βέβαια έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή ήταν η διεύρυνση. Οι χώρες που προσχώρησαν στη συνέχεια στην Ένωση είχαν λιγότερες δυνατότητες εφαρμογής ενό συντελεστών και δεσμεύονταν να σεβαστούν ε, τον κατάλογο που είχε προστατηθεί στο προσωρινό καθεστώς και στο μεταξύ αλλάξαμε άποψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του οριστικού καθεστώτος. Όχι πλέον προορισμό, όχι μάλλον καταγωγή που ήταν πριν, αλλά προορισμός πια. Αν κάποιο δηλαδή μπει στον κόπο να μετακινηθεί για να κάνει αγορέ σε ένα άλλο κράτο, υπόκειται στην νομοθεσία που ισχύει στο εν λόγω κράτο μέλο. Αν είναι μειωμένο συντελεστή, ακόμα καλύτερα για τον καταναλωτή. Δεν υπάρχει όμω πλέον η ανάγκη να εφαρμοστεί περιορισμός στο τι μπορεί να αποφεληθεί από τον μειωμένο συντελεστό. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα πια. Θα πούμε εμείς στην Πολωνία ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για τις πάνες, για παράδειγμα, όταν το κάνει η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δύο προβλήματα βλέπουμε εδώ. Το πρώτο. Ποιοι είμαστε εμείς που θα ορίζουμε στα κράτη-μέλη τι θα κάνουν, αν αυτό δεν είναι αναγκαίο και δεν έχει να κάνει με σεβασμό τη συνθήκη. Αυτό που θεωρήθηκε αντισυνταγματικό είναι το αντίθετο. Έχει γίνει γιατί ακριβώ πρέπει να τηρήσουμε το 113 άρθρο που λέει ότι πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση του κοινοτικού πλαισίου μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η εύρεθμη λειτουργία τη ενία αγορά και να αποφευχθούν οι στερευλώσει. Άρα χρειαζόταν να γίνει αυτό όταν είχαμε βάσει την ε, προέλευση και τώρα που έχουμε τον προορισμό χρειάζεται, όχι δεν χρειάζεται. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, κάποια περιθώρια φορολογικά. Ε, μία συνέπεια. Δεύτερο. Υπάρχει τώρα ε, εγγενής διάκριση, δεκτική μεταχείριση. Αν δεν αλλάξουν οι κανόνες πάβουν οι παρεκκλήσεις όταν άρχισε να ισχύει το οριστικό καθεστώς. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις. Και είναι και ανεδαφικό από πολιτικές πλευράς. Το θέμα είναι να κρατηθούν, να διατηρηθούν αυτές οι παρεκκλήσεις, αλλά να έχουν όλα τα άλλα κράτη της ίδιας ευκαιρίε και την ίδια δυνατότητα. Αυτό σημαίνει διάβρωση βάση βέβαια. Γι' αυτό και έχουμε βάλει μια πολύ σημαντική ασφαλιστική δίκλη για το σταθμισμένο ε, συντελεστή, που είναι 12% ε, το όριο του μειωμένου σταθμισμένου συντελεστή. Αν το κράτο μέλο έχει φορολογικά περιθώρια, φορολογικέ δυνατότητε για να χρησιμοποιήσει μειωμένου συντελεστέ ε, για να προωθήσει φορολογική πολιτική, κοινωνική, πολιτική, εισοδηματική, ανάπτυξιακή, αυτό είναι ελεύθερο να το κάνει. Εμείς απλά θέλουμε να καθοδηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το χωρίς να δίνουμε κίνητρα για αύξηση. Αλλά μια ελευθερία για να μπορεί να τον κατευθύνει όπως θέλει. Έξι λεπτά είναι πολλά είδη, ε, διακόπτει ο πρόεδρος. Έχουμε και άλλους τέσσερις στον κατάλογο. Μήπως μπορείτε τώρα να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι πολύ σωστά και έγκαιρα. Uh, Ευχαριστώ, αλλά υπερέβησαν οι προηγούμενοι ομιλητές μου ε, τέσσερα λεπτά το, λόγο, το χρόνο αγόρευσης, ενώ εγώ δεν τον είχα υπερβεί. Λοιπόν, η πρόταση για τον ε, πιστοποιημένο υποκείμενο σε φόρο. Να μην σας εξηγήσω, ε, αν δεν είστε ειδικοί, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Αλλά για να είμαι σύντομη. θέλουμε να πιάσουμε αυτού που εξαφανίζονται χωρί να έχουν πληρώσει φόρο. Και έχουμε βρει έναν τρόπο να το κάνουμε. Αν κάποιο ε, ε, πολλά ένα αγαθό ε, εκτό δεν φορολογείται και αυτό δημιουργεί την απάτη αυτή τη στιγμή. Αν αλλάξει ο κανόνα σημαίνει ότι θα πρέπει αμέσως να τα πιάσουμε αυτά τα χρήματα και να τα δώσουμε εκεί που πρέπει να πάνε. Είπατε εσείς ότι μπορεί τα κράτη-μέλη να φοβούνται ότι θα εισπράττονται από άλλον οι φόροι ή ε, για κάποιον άλλον. Εμείς έχουμε προτείνει αυτή τη βαθμιδόν προσέγγιση. Με αυτό τον CTP, τον πιστοποιημένο ε, φορολογούμενο, λέμε θα συνεχίσετε όσο διαρκεί αυτό το σύστημα αν το θέλετε, αλλά θέλουμε να πιάσουμε αυτούς που κεντρώνουν πιο πολύ να εξαφανιστούν με τα ε, λεφτά στην τσέπη. Να παραμείνει δηλαδή αυτή η κατάσταση που ισχύει στα κράτη-μέλη. Αλλά κλείνουν, βουλώνουν οι πιο μεγάλες τρύπε. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτή την λύση. Το δεύτερο ερώτημα ήταν η πρωτοβουλία από τα κρατη Εμείς για τις δύο χώρες που ζήτησαν να έχουν αυτό γενικευμένο σύστημα αντίστροφης χρέωσης, ε, τη συζητούμε την πρόταση, μάλλον συζητείται σε επίπεδο συμβουλίου. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Εμεί κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Θεωρούσαμε ότι τι προτάσει μα και με τη συνθήκη. Και τώρα το μπαλάκι είναι στο γηπέδο του συμβουλίου και πιστεύουμε ότι δεν είναι ασυμβίβαστα τα δύο μεταξύ του. Αλλά δεν θέλω να μπω σε νομικέ λεπτομέρειε, εκτό βέβαια αν μου το ζητήσετε. Υπήρχε και ένα τρίτο ερώτημα. Ε, ναι, έλεγα πόσο πιθανό είναι να τύχει επαρκούς υποστήριξη σε αυτή η πρόταση. Απάντηση. Όπως συμβαίνει και με οποιοδήποτε φορολογική πρόταση, θα χρειαστεί χρόνος. Αλλά βασιστήκαμε στην ε, αναπιθετική θηρίδα για τις υπηρεσίες και τώρα αφού πήγε καλά, το έχουμε βάλει σε όλε τι συναλλαγέ B2C εξ αποστάσεω. Έχει εγκριθεί η μονοπαθητική θηρίδα και θα πάει καλά. Στο Συμβούλιο εγκρίθηκε. Το μόνο που θα μένει θα είναι το B2B. Business to business. Είναι φυσικό. Και παραλαμβάνω, δεν μίλησα πιο πολύ από του επόμενου ομιλητέ την πρώτη φορά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανεί άλλο να σχολιάσει για τι ερωτήσει αυτέ. Σα παρακαλώ μου λάβετε υπόψη σα ότι έχουμε ακόμα τέσσερι ομιλητέ. Ευχαριστώ. Από ό,τι καταλάβω από την ερώτηση, ρωτάτε για την πρόταση για την αντιστροφή της χρέωσης. Να σας πω ότι το θέμα της έλλειψης εμπιστοσύνης και του εμπορευόμενου, ο οποίος δεν εντοπίζεται, είναι ένας τρόπος να επιτεθούμε στο πρόβλημα και αυτό συμβαίνει και στη διαδικασία της δημιουργίας εμπιστοσύνης, αλλά η πολιτική πίεση από κάποιους ο οποίος βρίσκεται υπεράνω της φορολογικής διοίκησης, ο οποίος λέει ότι αυτό το σύστημα πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Εάν υπάρξει τέτοια πολιτική πίεση, τότε θα υπάρξουν αλλαγές. Σίγουρα λοιπόν ε, πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη πολιτική πίεση για την εθνική ε, αντιστροφή της χρέωσης. Ρωτάτε αν θα αυξήσουμε τον κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση. Το όφελος είναι ότι όντως μπορεί να μειωθεί μία μορφή απάτης σε μία χώρα, με σαφή κίνδυνο όμως να εξάγουμε τον ίδιο τύπο απάτης στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και να το αντικαταστήσουμε και με ένα διαφορετικό κίνδυνο, διότι το προφίλ κινδύνου ε, από μια πληρωμή στην οποία συλλέγεται το τμήμα του ΦΠΑ ε, σταδιακά, όπου με ένα σύστημα το οποίο συλλέγει τα πάντα στο τέλος, ε, έχει τελείως διαφορετικούς κινδύνους. Μπορεί να δημιουργήσετε λοιπόν ένα νέο κίνδυνο και μια νέα πάτη χωρίς να το αντιληφθείτε. Το κατά πόσο θα πετύχει ή όχι να σας πω ότι καταρχήν το ΦΠΑ είναι ο πιο εύκολος φόρος στον κόσμο. Ε, εφαρμόζεται ένα συντελεστή σε μια συναλλαγή, αλλά καταφέραμε να το ε, κάνουμε πολύ σύνθετο. Ευχαριστώ, πολύ σαφές και απόλυτα αντιληπτό. Περνάμε στον ε, εισηγητή για τον πιστοποιημένο υποκείμενο στο φόρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η τελική παρατήρηση. Καταρχάς, ε, νομίζω ότι πολλά από τα θέματα ε, που συζητήθηκαν είναι και πράγματα που έχουμε συζητήσει στο θέμα που απασχολεί εμένα στην έκθεσή μου και φυσικά όλος λόγος ε, γίνεται για να έχουμε ένα απλό σύστημα ώστε να προλάβουμε και να καταπολεμήσουμε τη διασυνοριακή απάτη και να δώσουμε και μια όθηση στο εμπόριο. Αυτά είναι τα βασικά. Ε, να μην ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί υπάρχουν πολλέ ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ. Ο Κρίστιαν, για παράδειγμα, νομίζω ότι αναφέρθηκε πολύ στην έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών και στο γεγονό ότι δεν λαμβάνονται σωστέ πληροφορίε, δεν ε, καταλαβαίνει ένα τον άλλον κλπ. Μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε λίγο περισσότερα για το πώ μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχετε κάποιες προτάσεις, αναφερθήκατε σε κάτι, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνης και συνεργασίας των κρατών μελών στα θέματα αυτά. Και επίσης, ο Γκέρχαρτ, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε και δύο λόγια παραπάνω για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόσκομα. Το αναφέρατε ε, ακροθυγώς αυτό το νέο σύστημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σε σχέση, σε σύγκριση και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Μήπως υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη να ασχολούμαστε με το θέμα. Ευχαριστώ. Να δώσω πρώτα λοιπόν το λόγο στο Γκέρχαρτ γιατί είναι ο πρώτος στον οποίο απευθύνθηκε το ερώτημα και μετά να απαντήσει κάποιος από το πάνελ. Εκτός και αν έχετε κάποια προτίμηση. Ο Κρίστιαν πρώτα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός και συγκεκριμένο. Για την, για την δημιουργία εμπιστοσύνη. Πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνη, Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πάντα κρεμεί. Η αρχική πρόταση για μια ομοφθητική θηρίδα είχε ένα χαρακτηριστικό που έλεγε ότι υπάρχει κάποια μορφή πληρωμή από το κράτο μέλο για να γίνει ο έλεγχο, ο οποίο προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει υπερβολική απερβάρυνση για να γίνονται φορολογικέ διαδικασίε εκ μέρου άλλου κράτου μέλου. Το κατά πόσο είναι καλή αρχή ή όχι, νομίζω δεν έχει σημασία γιατί τα κράτη-μέλη είπαν δεν θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά η συνεργασία, η μονοαπευθυντική φυρίδα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τώρα για το B2C είναι το πρώτο βήμα ε, στο οποίο προσπαθούμε να συλλέξουμε ΦΠΑ εκ μέρου άλλων. Αυτό σημαίνει δημιουργία εμπιστοσύνη. Θα καθυστερήσει λίγο, αλλά στην ουσία είναι ένα από του καλύτερου καταλήτε για να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνη. Επίση, να βρεθούν και κάποιοι τρόποι να συνεργαστούν Εάν συναντηθούν ε, ως ε, ε, φοροσυλλέκτης και ως φορολογική υπηρεσία κάποια από άλλα κράτη-μέλη, τότε ξέρεις πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, μπορείτε να συνεργαστείτε. Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε, για παράδειγμα, ένα συνοριακό έλεγχο. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε ένα, δύο, τρει μήνες να λάβουμε απάντηση. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα δίνεται μια σύντομη απάντηση, διότι ο απατεώνας ε, κρύβεται πίσω από τα σύνθετα πράγματα και κρύβεται πίσω από την έλλειψη συνεργασίας. Εάν χρειάζεται λοιπόν τρεις μήνες για να γίνει ε, τη χάσαμε την απάτη. Όσον αφορά την έλλειψη ενημέρωσης. Έχουμε τονίσει και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει συμπεριλάβει και αυτό στη δικτυακή πύλη για τις πληροφορίες ΦΠΑ. Στην ουσία θα μπορούσατε να αναρωτηθείτε γιατί ένα κράτος μέλος να μην θέλει να αναρτήσει δημοσίω τον ε, εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ σε μια δικτυακή πύλη ΦΠΑ. Γιατί να μην το εκμεταλλευτούν από αυτό και να πούνε βεβαίω θέλουμε να διευκολύνουμε τη συμμόρφωση. Και πρέπει να σα πω εγώ προσωπικά δεν βρίσκω απάντηση αλλά νομίζω ότι το κόστος ε, διατήρησης της πληροφορίας είναι σημαντικό, αλλά θα έπρεπε να είναι προς το συμφέρον όλων να αναρτώνται αυτές οι πληροφορίες και να είναι εύκολες, προσβάσιμες και αξιόπιστες. Δεν μπορείς να ζητήσει από έναν έμπορο ο οποίος δεν είναι ειδικό σου επί α ο ίδιος να πρέπει να βρει και να, ή να συμβουλευτεί κάποιον άλλον για το πώς έχει ο συντελεστής, πώς ε, γίνεται καταχώρηση και πώς θα λάβει επιστροφή ΦΠΑ. Δεν γίνεται αυτό στο σημερινό κόσμο. Ο Γκέχαρτ. Για, από πλευρά τη μικρομεσαία επιχείρηση έχουμε δύο προβλήματα με την πρόταση για τον πιστοποιημένο υποκείμενο στο φόρο. Καταρχά, αν είσαι προμηθευτή, στο μέλλον δεν θα πρέπει να γίνει μόνο διάκραση εάν ο πελάτη σου στο εξωτερικό είναι καταναλωτή ή κάποια άλλη επιχείρηση, αλλά θα πρέπει να δει αν είναι ε, πιστοποιημένο στο φόρο ή όχι. Άρα, χρειάζεσαι ένα σύστημα πληροφοριών το οποίο θα λειτουργεί απόλυτα, θα είναι αξιόπιστο και θα παρέχει τις πληροφορίες αυτόματα, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλιώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα σωστά από νομική σκοπιάς. Δεύτερον, αν είσαι ο παραλήπτης ε, και αν έχουμε προμήθεια B2B από επιχείρηση σε επιχείρηση και δεν μπορείς να πάρεις πιστοποιητικό πιστοποιημένο πιστοποιημένος υπόχρεωστο θόρο, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ σύνθετες ιδέε και θα είναι πολύ δαπανερό για μικρές επιχειρήσεις να κάνουν κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να καταβάλεις ΦΠΑ για την προμήθειά σου και ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ΦΠΑ και ο άλλος που έχει πάρει την πιστοποίηση δεν θα παίρνει ΦΠΑ και αυτό φυσικά δημιουργεί πρόβλημα συμμόρφωσης. μπορούμε να υποστηρίξουμε το σύστημα του, υπόχρεου, του πιστοποιημένου υπόχρεου στο φόρο εάν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση έχει εύκολη πρόσβαση με χαμηλό κόστος ευθύ εξ αρχή στο νέο σύστημα. Αλλιώ θα δημιουργηθεί πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Δεδομένου του ότι έχουμε τρεις ε, ομιλητές ακόμα ε, και ε, επειδή αρχίσαμε πιο αργά ας προσθέσουμε μερικά λεπτά ακόμα διότι έχω πληροφορίες ότι το επόμενο θέμα θα τελειώσει πιο γρήγορα. Ο κύριος Ζήλε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ε, πολλές συζητήσεις ε, στο Κοινοβούλιο σχετικά ε, με το συγκεκριμένο σύστημα. Όμως η δική μου ανησυχία είναι λίγο πιο γενική. Νιώθω ότι η καθηγήτρια Φερία έκανε μερικά πολύ καλά σχόλια ε, όσον αφορά την πρόταση. Όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις μας ε, δεν μπορούσα να εντοπίσω τόσο έντονα μια τέτοια κριτική προσέγγιση όμως αν την κατάλαβα καλά είπε ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι αντισυνταγματική ε, και οικονομικά ε, λαθασμένη. Ε, οκ, δεν το αποκλείω. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε πια είναι η εναλλακτική. Διότι πιστεύω ότι πολύ έργο έχει δαπανηθεί για αυτήν την πρόταση, οπότε είναι έκπληξη για μένα αυτός, αυτή η αυστηρή κριτική όμως ε, ποιες είναι οι που θα προτείνατε ε, και στο πλαίσιο των δύο λεπτών που έχω θα ήθελα επίσης ε, να τονίσω και κάτι ακόμα. Ο ΦΠΑ δεν είναι απλά ένας ξένος παίκτη εντός του οικονομικού κόσμου είναι διασυνδεδεμένος με πολλά ζητήματα φορολόγησης ε, και υπάρχουν χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν ένα υψηλό ε, ΦΠΑ για να μπορέσουν ε, να, σε αντάλλαγμα των επιδομάτων και των βοηθειών που προσφέρουν. Όμως το βασικό μου ερώτημα, όπως και να έχει, αφορά την εναλλακτική στην πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το ερώτημα ήταν για την καθηγήτρια Λαφέρια. Όλα τα σχόλια τα οποία έκανα πάνω στην ε, πρόταση αναπτύσσονται αναλυτικά στα ε, έγγραφα τα οποία προώθησα στην Επιτροπή ε, και τα όσα δήλωσα εδώ πέρα αποτελούν τα συμπεράσματα, τα ε, επιχειρήματα είναι τόσο, έχουν τόσο πολιτική όσο και οικονομική ε, βάση και τα αναλύω στα, στα, στις εργασίες μου. Καταλαβαίνω ότι πολιτικά είναι δύσκολο όλο αυτό, όμως το θέμα είναι ότι ίσως να κάνουμε χειρότερη την κατάσταση από ό,τι είναι. Η κατάσταση δεν είναι ιδανική, δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή. Το ευρωπαϊκό σύστημα FPI είναι αναχρονισμένο, διουργεί σε προβλήματα στον ανταγωνισμό, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για τι μικρέ και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αποτελεί εμπόδιο στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Όλα αυτά ναι ισχύουν, όμω, ο φόβο μου είναι ότι η πρόταση όπω είναι θα κάνει τα θέματα αυτά ακόμα χειρότερα, διότι αν έχουμε περισσότερη διαφοροποίηση και στρέβλωση τη βάση, τότε η κατάσταση θα είναι ακόμα χειρότερη και ο φόβο μου αφορά και τι ε, συνέπειε όσον αφορά τα έσοδα. Εάν συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε δεχόμαστε τη διάβρωση της βάσης ακόμα και αν υπάρχει ένα όριο όπως είπε η Κομισιόν Εάν συνεχίσουμε αυτό το μονοπάτι διάβρωσης της βάσης, τότε θα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ελλείμματος εσόδων και είτε θα πρέπει να, να μειώσουμε τις ε, δημόσιες παροχές ή να βρούμε τα χρήματα από αλλού. Το ΦΠΑ είναι ένας καλός τρόπος εσόδων, καλή πηγή εσόδων για να παρέχουμε τις, τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Όμως ε, φοβάμαι ότι ε, δεν θα βρίσκουμε τα χρήματα και δεν βλέπω την όρεξη αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά δεν είμαι πολιτικός, αλλά με βάση τα όσα βλέπω να συμβαίνουν στην Ευρώπη ως μάρτυρας, ως πολιτικός συμμετέχων, δεν βλέπω την όρεξη για την μείωση των ε, κρατικών παροχών. Αυτή είναι η φόβη μου λοιπόν Πρώτον, λοιπόν, ότι θα αποτρέψει, θα θέσει εμπόδια στο ευρωπαϊκό, ε, στο ευρωπαϊκό εμπόριο, θα δημιουργήσει πιο έντονη στρέβλωση και επίσης θα χάσουμε έσοδα τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν σε δημόσιες υπηρεσίες. Δεν βλέπω άλλο τρόπο λοιπόν να το επαναρθώσουμε αυτό και είναι σημαντικό για μένα ε, το να τονίσω δεν βλέπω το λόγο να κάνουμε κάτι τέτοιο για ποιο λόγο να διαβρώσουμε τη βάση ΦΠΑ βλέπω καλούς λόγους για να μεγαλώσουμε τη βάση αλλά δεν βλέπω καλούς λόγους είτε από πολιτικής, νομικής ή οικονομικής άποψης να διαβρώσουμε τη βάση και γι' αυτό τον λόγο ασκώ κριτική στην πρόταση. Ε, τα ε, papers τα οποία έχω γράψει ε, μπαίνουν σε λεπτομέρειες για όλο αυτό και θα χαρώ να συζητήσω με οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής ξεχωριστά εκτός της αίθουσας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι η κυρία Λεζιόν θέλει επίσης να απαντήσει. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Συμφωνώ ότι ε, οι ε, καλύτερες ε, πρακτικές αφορούν την βάση και εδώ κινούμαστε σε, προς ένα οριστικό καθεστώς ώστε οι χώρες να έχουν την απόλυτη ελευθερία. Υπάρχει ένας περιορισμός σχετικά με το πού μπορείς να κινηθείς. Όλο αυτό δεν είναι ατελείωτο συμφωνώ ότι έχετε ανησυχίες, ίσως όμως ταυτόχρονα υπάρχουν ε, εμπόδια στα ελλείμματα και στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Υπάρχει ο μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και παρόλο που είμαι υπέρ και παρόλο ε, που διδάσκω ε, φορολογικό δίκαιο των επιχειρήσεων, πιστεύω ότι η πρόταση θα πρέπει να βασίζεται στην απόφαση του κρατούς μέλους και υπάρχει όριο σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν. Και ένα τελευταίο σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω όσον αφορά τα ε, ποσοστά είναι ότι αν έχουμε διαφορετικά ποσοστά ε, στις χώρες ε, θα πρέπει να αναλογιστούμε ίσως να να χρησιμοποιούσουμε όλες αυτές τις ε, στατιστικές που χρησιμοποιούνται ε, μονάχα για τα προϊόντα τα οποία θα πρέπει να έχουν ε, βασική κατηγοριοποίηση αλλά να το κάνουμε αυτό και σε άλλα ποσοστά τα οποία ορίζονται από τις χώρες διότι αν αρχίζουμε να εμπορευόμαστε σε διαφορετική δικαιοδοσία ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη ταξινόμηση ε, η οποία θα επιτρέπει και την αυτοματοποίηση για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ακολουθεί ο κύριος Λούκα από το ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. έχω ερωτήματα από επί της αρχής. Ε, αν ακολουθήσουμε ε, την ε, πρόταση της Κομισιόν και πάμε στην αρχή της χώρας στόχος, τότε ο καλύτερος τρόπος θα είναι με την αντίστροφη μέθοδο, διότι εάν θεωρήσουμε ότι ο φόρος ε, θα επιβάλλεται εκεί που υπάρχει ο τελικός καταναλωτής, τότε ή για μένα είναι παράλογο ε, να το κάνουμε αυτό κατά τη διάρκεια της αλυσίδας. Οπότε η διαδικασία θα πρέπει να είναι αντιστρωμένη. Και επίσης το ερώτημα ε, όσον αφορά τον έμπιστο, την καταγραφή του έμπιστου εμπόρου. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας εξηγήσετε πού θα ήταν ο κίνδυνος αν έχουμε αυτό το σύστημα καταγραφής έμπιστου ε, εμπόρου ε, διότι το πρόβλημα νέων δυνατοτήτων ε, γίνεται πιο έντονο αν έχουμε αυτό το σύστημα. Ίσως όμως και να κάνω λάθος. Το τελευταίο μου ερώτημα αφορά τη διάβρωση της βάσης ε, που ε, τονίσατε εσείς. Δεν το εντοπίζω που ακριβώς βρίσκεται και θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε διότι αυτό το οποίο είπατε είναι ότι θα υπάρχει μια τάση ε, προς ε, μειωμένα ε, ποσοστά ΦΠΑ στο σύστημα, όμως αυτό διαφέρει από τη βάση. Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα λεπτάκι πρώτα να θέσω την ερώτησή μου. Δεν βλέπω λοιπόν που υπάρχει αυτή η διάβρωση. Επίσης δεν κατανόησα τον μηχανισμό ο οποίος θα οδηγήσει σε πιο μειωμένα ποσοστά από τα ίδια υπάρχοντα. Είναι δύο θέματα λοιπόν, αφορά τη βάση, αφορά τα ποσοστά ε, και επίσης ε, οι χώρες οι οποίες ε, αυξάνουν το ΦΠΑ θα έχουν ένα σύστημα με μειωμένα έσοδα. Δεν βλέπω τι εννοείται με όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν κάποια ερωτήματα. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει. Ας ξεκινήσουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά με την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το ε, ΦΠΑ λειτουργεί με μεμονωμένες πληρωμές. Αυτή τη στιγμή το σύστημα το οποίο έχουμε είναι μεταβατικό ε, καθεστώς και είναι de facto ένα τέτοιο σύστημα όσον αφορά το διασυνορικό B2B. Και εκεί ξεκινά το πρόβλημα διότι Ε, διότι αλλάζει όλους, ε, όλο το σύστημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όταν ε, μπαίνουμε στην μαύρη αγορά χάνουμε τα πάντα και ξεκινώντας με αυτές τις πληρωμές αν έχουμε ακόμα και ένα κομμάτι της αλυσίδας το οποίο χάνεται χάνουμε μονάχα αυτό το κομμάτι του ΦΠΑ και όχι ολόκληρο. Έτσι λοιπόν από την μία πλευρά υπάρχει αυτό το γενικό πρόβλημα όσον αφορά τον ΦΠΑ σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο πράγμα ε, το σύστημα αυτό διεθνώς και ε, στο εσωτερικό των χωρών το γεγονός ε, δηλαδή ότι η προμήθεια φορολογείται το γεγονός ότι ο φόρος αυτός υπάρχει είναι επειδή δεν έχουμε ένα ομοσπονδιακό σύστημα έχουμε διαφορετικές φορολογικές αρχές όμως στη μάχη κατά της απάτης και την απλοποίηση του συστήματος ε, θα ε, πρέπει, ε, είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή αποτελεί μια καλύτερη εναλλακτική. Όσον αφορά την καταγραφή του έμπιστου εμπόρου, Πού είναι το πρόβλημα με την αντιστροφή της χρέωσης, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε όλους απαντά και τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους. Δεν μπορούμε να κινηθούμε μονάχα για ένα ε, κομμάτι. Είναι μια ε, πολυπλοκότητα που δεν χρειάζεται. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ. Μπορούμε να το δούμε αυτό στην αξιολόγηση αντιτύπου, να δούμε τις εναλλακτικέ Ευχαριστώ. Ε, φαίνεται ότι η καθηγήτρια Λεφιέρα θέλει να απαντήσει. Θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπε η Έλενα, η Κομισιόν, θέλω να πω, για την τροφή της χρέωσης. Η έρευνα δείχνει ότι όταν ε, ότι ο ΦΠΑ έχει ε, υπερτερή αν θέλετε, έχει προβάδισμα σε ό,τι αφορά την απάτη. και είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος από ότι όταν έχουμε ένα μόνο τμήμα της παραγωγής που μας απασχολεί. Και η αναφορά από τρίτο, η αναφορά της συναλλαγής από τρίτον επίσης επηρεάζει και αυξάνει τις ε, εκθέσεις και τις αναφορές πωλήσεων και όχι το αντίθετο σε ό,τι αφορά του συντελεστές ΦΠΑ. Η διάβρωση της βάσης είναι τεχνικός όρος για οτιδήποτε δεν υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Η υποθετική βάση ΦΠΑ είναι οτιδήποτε καταναλώνεται σε μια δεδομένη χώρα και πάγεται, υπόκειται στον κανονικό συντελεστή. Οτιδήποτε παρεκκλίνει από αυτό, από την πλευρά των δημόσιων οικονομικών, θεωρείται φορολογική δαπάνη, εφαρμόζεται μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ από ό,τι θα ίσχυε κανονικά. Από εκεί προέρχεται η διάβρωση βάση σε ό,τι αφορά τις πιέσεις, γιατί τα κράτη-μέλη το κάνουν. Διότι έχουμε δει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη, όχι μόνο μία χώρα. Θα μπορούσα να σας δώσω πολλά παραδείγματα. Στο Ενωμένο Βασίλειο, τα, τα, ε, τα βιβλία, τα παπούτσια σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία έχουμε άλλο θέμα με άλλο είδος. Και Πολλέ φορές το κόστος από τη μέση του συντελεστή είναι τεράστιο. Αν οι ομάδες πίεσης αντιληφθούν ότι υπάρχει δυνατότητα για χαμηλότερου συντελεστέ, θα ασκήσουν περισσότερη πίεση προς αυτό. Έτσι βλέπω εγώ να πηγαίνει. Όχι να αυξάνονται λόγω πολιτικής πίστης, αλλά μειώνονται. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να απαντήσει από το πάνελ, γιατί κοντεύμα ολοκληρώσουμε εσείς. Ναι κύριε Λεζέν, συμφωνώ. Μέσα στην ίδια αλυσίδα να έχουμε ίσπραξη φόρων και αντίστροφη της χρέωσης. Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, αλλά λέω γι' αυτό ακριβώ χρειάζεται αυτή η μονοπαθητική θύρη, για την ίσπραξη. Και θέλουμε να γίνει η χρέωση και δεν θέλουμε να γίνει με κάποιον τρίτο Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε το σύστημα εμπιστού εμπόρου μέσω της καταχώρησης. Ανεξαρτήτως του κατά πόσον γίνεται αντιστροφή της χρέωσης. Τι ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο συστήματα. Υπάρχουν δυνατότητες αρμπιτράζ. Όχι από νόμιμους εμπόρους, αλλά από εγκληματίε που εμείς δεν τους θέλουμε στο σύστημα. Ευχαριστώ Άλλους ένας. Θα περιπλέξω μάλλον τα πράγματα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. για να έχουμε ισορροπία. Με χρέο του ΦΠΑ θα μπορούσε κανεί να πει ότι αλλά έχουμε ένα απλό σύστημα χωρίς ε, να λείπει κάποιο κρίκο. Και υπάρχουν τρισεκατομμύρια καθάριστου ΦΠΑ που δεν ε, είναι αυτό που παίρνουμε ουσιαστικά, αλλά αυτό που πρέπει να επιστραφεί, να εισπραχθεί κτλ. Είναι τεράστιο το ποσό που πρέπει να επιστραφεί διασυνοριακά αν χρειαστεί. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είμαστε υπέρ μεθόδων απλούστευσης. Όπως έχει όμως η πρόταση αυτή τη στιγμή, δεν πιστεύουμε ότι είναι η σωστή απάντηση στο ποιημένο υποκείμενο στο φόρο, διότι δεν ξέρουν πάνω σε τι ε, θα εφαρμοστεί το σύστημα. Σε κάποιες ε, ομαδικές ε, πωλήσει. Τι ακριβώς αυτά αφορά αυτό το σύστημα. Για να το απαντήσουμε το ερώτημα πρέπει να ξέρουμε πόσο πολύπλοκο είναι αυτό και τι απλουστεύσει θα χρειαστεί το σύστημα. Μπορεί να μην είναι αυτή η ιδανική απάντηση. Ειλικρινά όμως, το να συζητάμε αυτό το πιστοποιημένο πώς να ξέρουμε τι συναλλάσσεται αυτός ο άνθρωπος, η φορέας είναι λίγο δύσκολο. Thank you very Σας ευχαριστώ. Η Μόλι Σκοτ Κέιτο δυστυχώς έφυγε. Επειδή καθυστερούσαμε εδώ, τελείωσε ο γύρος ερωταπαντήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και δι' τους προσκεκλημένους. Βέβαια αυτή ήταν η απαρχή μόνο της συζήτησης. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο κοινοβούλιο αυτή η πρόταση. Φαντάζομαι θα έχουμε και άλλες συζητήσεις ε, πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που θα μας εμπλουτίσουν. Δεν σταματάει εδώ λοιπόν αυτή η συζήτηση. Απλά αναβάλλεται για κάποια προσεχή συνεδρίαση. Και εμείς σίγουρα στο μέλλον θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για μια ακόμη φορά για την καθυστέρηση που οφείλεται στο ότι η προηγούμενη συνεδρίαση κράτησε περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της Μέσης Διάταξης, το υπάρχουν 13. Να γίνει μια αλλαγή φρουράς εδώ. Ε, εγκαταλείπουν την αίθουσα οι προσκεκριμένους, ο οποίος ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. This is updated. I don't know whether you have this already. Maybe there are some more names. No, it's the same. It's the same. So. And the timeline is on the back, you know, because we agreed that yesterday. Yeah, yeah, I have it also. I have it. So, dear colleagues, let me start point number seven. Από τη περάσουμε στο σημείο 13, ένα σημαντικό σημείο, γενικό περιπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, όλα τα τμήματα. Έχουμε τον εισηγητή για τον προπολογισμό τον κύριο Ντανέλε Βιώτη από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Συγγνώμη που περιμένετε 10 λεπτά κύριε Βιώτη. Θα συμμετάσχετε στην συνάντηση και θα κάνετε μια γενική εισαγωγή της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού. Θα μιλήσει έπειτα ο εισηγητής ε, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από την ΕΚΟΝ. Όπως προβλέπουν οι διαδικασίες, θα έχουμε δύο ουσιαστικά σκέλη διαδικασίας γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ για τον προπολογισμό θα υποβληθεί στην καθήλυνα αρμόδια την Επιτροπή Προπολογισμών ε, που θα δίνει τα πολιτικά μηνύματα και τι ε, πολιτικέ τροπολογίε για τροποποίηση των αριθμητικών στοιχείων που θα γίνει ξεχωριστά. Η Κομισιόν στις 23 Μαΐου θα καταθέσει αυτό το προσχέδιο. Δηλαδή συστάμε για κάτι που ακόμη δεν έχει ε, διατεθεί. Καταρχά να δώσω το λόγο στον εισηγητή Επιτροπή Προπολογισμών, τον κύριο Βιώτη. Πέντε λεπτά θα έχετε για να κάνετε την εισαγωγή και έπειτα θα περάσουμε στους συζητητές από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χίλια ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους της Επιτροπής ε, που με φιλοξενούν εδώ σήμερα, διότι ε, παρά το γεγονός ότι μας πιέζει ο χρόνος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται ένας ε, εις βάθος διάλογος με όλους τις επιτροπές και φυσικά την επιτροπή σας. Και θα ήθελα να κάνω αυτό το γύρο των επιτροπών και να ακούσω και την άποψή σας. Και από πλευράς μεθοδολογίας, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, διότι η πρόθεσή μου, όπως και όλων των υπολείπων προηγούμενων εισηγητών, είναι στο μέτρο που μπορούμε να σας παρουσιάσω κάτι το οποίο θα χαίρει τη ευχαρίστηση του Κοινοβουλίου και να έχουμε μια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια στεναρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν θα πρέπει ε, να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διαπραγματευτούμε. Ε, τα θέματα τα οποία ε, έχω εντοπίσει και εδώ περιμένω τις προτάσεις σας και την άποψή σας τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον ετούσιο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν καταρχάς και την ε, μεταρρύθμιση και τα τομεακά προγράμματα και τη μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας. EBA, ΕΣΜΑ, e IPOP ε, και τη μεταρρύθμισή τους, ε, τα οποία φυσικά θα έχουν και αντίκτυπο στον προπολογισμό, μέσω της πρότασης ε, του κεντρικού αντισυμβαλόμενου και του CCP. Ε, υπάρχουν θέματα υποπτίας που αφορούν και τα CCP τρίτων χωρών. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει επιπλέον κόστος, το οποίο θα ε, θα τα παίρνουμε από το 2019 από τις ποσοστώσεις του CCP, αλλά χρειάζεται και ένα ε, τμήμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού για να γεφυρώσει το 2018 και το 2019 για τους πρώτους 12 μήνες ε, των, ε, ε των συναλλαγών πριν τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα των ποσοστώσεων. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη, το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει με τον προπολογισμό να δώσουμε μια γέφυρα μέχρι το 2019. Και μετά υπάρχει πρόταση για τα πανευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά χρηματοδοτικά συστήματα σε ιδιωτικό επίπεδο, το οποίο αφορά ε, την ε, ε, καταχώρηση και την εφαρμογή των οργανισμών συντάξεων που έχουν καταγραφεί. Θα γίνουν επί τη βάση 60-40 με τα κράτη-μέλη. Η συμβολή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι το 40% και θα είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για το 2019 και το 2020. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά ε, στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν και την Επιτροπή ΕΚΟΝ για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019. Αλλά όπως σας είπα, είμαι εδώ για να ακούσω φυσικά και τις δικές σας τις προτάσεις και τις δικές σας απόψεις και ό,τι έχετε να μου πείτε προκειμένου να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο για τον προπολογισμό του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιώτη να πάρει το λόγο υποφαινόμενος, γιατί είμαι και εισηγητής ε, για την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Καταρχάς να σας πω, όπως ε, γνωρίζετε, συζητούμε την πρόταση η οποία ακόμα δεν υπάρχει. Επομένως θα ήθελα να σας πω λίγο ε, κάποια προκαταρκτικά σχόλια και κάποιες απόψεις όσον αφορά τη γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ για τον προπολογισμό. Καταρχάς, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλά και παγκοσμίω, πρέπει να λάβουμε υπόψη και οικονομικά θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και ποιε είναι οι βασικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω την άποψη ότι στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο υπάρχουν κάποιε πολύ ισχυρέ προτεραιότητε, όπω τα θέματα ασφάλεια και άμυνα, και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και αντίστοιχη χρηματοδότηση στον προπολογισμό για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι γραμμέ προπολογισμού που είναι τη εμπειρογνωμοσύνη τη ΕΚΟΝ θα είναι απόλυτα ισορροπημένοι και αρμόδιοι οργανισμοί ε, και οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν και να μην υπάρχουν περιττέ πιέσει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Οι αλλαγέ μπορούν να γίνουν αποτελεσματικά και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνον τότε και είναι αιτιολογημένο θα μπορέσουμε να εξετάσουμε και τη χρηματοδότηση. Όσον αφορά τη δομή του προηγούμενου προπολογισμού, μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν την ΕΚΟΝ είναι ε, το σχέδιο Juncker για το οποίο πρέπει να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και το επόμενο θέμα το οποίο είναι απόλυτα σαφές είναι οι αυξημένες απαιτήσει ε, για την, ε, τον αυξημένο προπολογισμό των ε, ESA. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα υπάρχει και αυξημένη ευθύνη αυτών των υπηρεσιών. Αν δούμε πιο προσεκτικά τις γραμμέ προπολογισμού, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν επικαλύψεις ε, και διπλά στοιχεία. Ε, θα πρέπει να δούμε τον προπολογισμό ώστε να μην υπάρχουν περιττές επικαλύψεις και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η άξιση των ε, του προπολογισμού για κάποια θέματα θα συνοδεύεται και από αντίστοιχη μείωση κάπου αλλού, γιατί είναι μπλοκαρισμένα στι δυνατότητε του προπολογισμού. Θέλω συμβολή από όλου του σκιώδει εγγελτέ και από τα ε, μέλη της ΕΚΟΝ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην πολύ σημαντική δουλειά των συναδέλφων στην Επιτροπή Προπολογισμών. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τώρα εδώ με τις απόψεις μου, διότι δεν ε, είναι εδώ όλοι οι σκιώδεις συγητές. Ε, να δώσω το λόγο βέβαια στην κυρία Μπερές για να μιλήσει για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από, εκ μέρου τη Σιμώνα Μποναφέ, η οποία δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Να ευχαριστήσω το Γενικό Εισηγητή του Προπολογισμού, της Επιτροπής προπολογισμό. Νομίζω ότι πολύ καλά ε, κατάλαβε ποια είναι τα στοιχεία που απασχολούν την Επιτροπή μας ε, για το 2019, για τον προπολογισμό. Να υπενθυμίσω ότι πέρσι υπήρχε σταθεροποίηση των προπολογισμών των ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών και οργανισμών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το περιεχόμενο. Δεύτερον, εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν λόγω του Brexit, διότι είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι άμεσα προφανές, αλλά έχει ήδη ένα πολύ σημαντικό αντίκτυπο και το βλέπουμε όταν έχουμε άμεση επαφή ε, με τις τρεις υπηρεσίες ε, και την υπηρεσία για τις τράπεζες ε, και για τις ασφάλειες και τις συντάξεις και για τις, κινητές, για ακίνητες αξίες. θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό ε, καθεστώ όσον αφορά τις συντάξεις. Βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει πολλή δουλειά για τις υπηρεσίες και νομίζω ότι υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν αναφέρθηκε, αλλά μπορεί να δεν πρόσεχα κιόλα. Είναι ο αντίκτυπος της μετεγκατάστασης της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τραπεζών είχαμε έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά νομίζω του χρόνου θα έχουμε την πλήρη δραστηριότητα για να λάβουμε υπόψη και τη μετεγκατάσταση της υπηρεσίας. Έχουμε δηλαδή μια παράλληλη διαδικασία. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε σύγκριση και να δούμε τι γίνεται και με τον ε, οργανισμό φαρμάκων, αλλά είναι και ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Όλα αυτά βέβαια εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αν όλα πάνε καλά, δεν ξέρω αν θα πάνε καλά, μπορεί να υπάρχει ένας νέος τρόπος χρηματοδότησης των υπηρεσιών αυτών και να εφαρμοστεί, διότι όπως γνωρίζετε γίνεται αναθεώρηση των εποπτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή και αφορά και τις τρεις υπηρεσίες και στην οποία προβλέπεται, τουλάχιστον αυτό έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρχει μεγαλύτερη συμβολή από τους παράγοντες της αγοράς για τους συγκεκριμένου οργανισμούς. Και επομένως ο ευρωπαϊκός προπολογισμός θα πρέπει να περιορίσει τη συμβολή του ε, σε ένα μέγιστο του 40% των προπολογισμών αυτών των υπηρεσιών. Δεν ξέρω αν αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2019. Μπορεί να μου πείτε ότι ίσως όχι, αλλά ε, φαντάζομαι ότι θα αλλάξει η χρηματοδότηση για αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω. Πέραν των όσων ε, είχε πει η κυρία Σιμώνα Μπεναφέ, η οποία βέβαια όταν έρθει θα σας πει πολύ περισσότερα γιατί έχει εμπειρογνωμοσύνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μουσκιώδησα από το ECR. Είναι εδώ, όχι, κυρία Σουίμπεν, δεν είναι εδώ, το κύριος Λουκε θέλει να σχολιάσει από την άλλη. Και Γέζεκ δεν θέλετε να σχολιάσετε εσεί και του πράσινου. Είναι ο Σφεν Γκίγκολ και οι Δεν υπάρχει όμω ούτε ένα πράσινο στην αίθουσα. Απ' την ΚΟΥ υπάρχει κανεί εδώ. Yeah, is just money, you know. Ε, για λεφτά μιλάμε, γι' αυτό δεν είναι κανείς εδώ. Υπάρχει κάποιο που θέλει να πει κάτι από οποιαδήποτε ομάδα ουδής. Είμαστε πολύ καλά σε ό,τι αφορά το χρόνο. Στο πλαίσιο τη διαδικασίας κάτι διάει, Όχι. Ο καλεσμένος μας. Μήπως θέλει να απαντήσει ο κ. Βιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη συμβολή σας και να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο Μπερέσου για την ε, ε, πολύ σημαντική συμβολή της. Ε, προφανώς και τα σημείωσα όλα και είδα και τα στοιχεία τα οποία μου αναφέρετε. Θα ήθελα εδώ να κάνω δύο παρατηρήσεις ε, κλείνοντας για τα όσα μου είπατε και φυσικά θα περιμένουμε και τον προπολογισμό, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, γιατί ούτως ή άλλως προς το παρόν συζητάμε για το τίποτα, γιατί δεν έχουμε ε, προσχέδιο προπολογισμού της Επιτροπής, ε, θα μας το στείλουν τέλη Μαΐου. Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας πολύ σωστά είπατε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποιους πόρους από αυτού. Εμείς συμφωνούμε ότι η ασφάλεια και η έμεινα, ιδιαίτερα το νέο σχέδιο για την άμυνα, πρέπει να έχουν και αντίστοιχους πόρους, αλλά αυτό όχι εις βάρος ε, ε, υφιστάμενων προγραμμάτων. Ε, όταν η αρχή που διέπει λοιπόν ε, ε, ε, την Επιτροπή Προπολογισμών και γενικότερα το Κοινοβούλιο είναι ότι όταν έχουμε νέες δαπάνες τότε θα πρέπει να υπάρχουν και νέα έσοδα. Όταν ζητάμε νέα προγράμματα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να φέρουμε κονδύλια από άλλα προγράμματα τα οποία είναι στα σκαρδιά γιατί φυσικά αυτό είναι εις βάρος και των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ιδίως των μικρομεσαίων και ούτω καθεξής. Μία ακόμα μικρή σκέψη, επειδή συγκέντρωσα εδώ όλα αυτά που μου είπατε όσον αφορά τα καθήκοντα των υπηρεσιών και των οργανισμών και σε αυτή την περίπτωση εμείς εδώ και χρόνια είμαστε μάρτυρες ε, της μείωσης κατά 5% του προσωπικού όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των θεσμικών οργάνων αλλά όταν αναθέτουμε νέα καθήκοντα και νέε αρμοδιότητε στι υπηρεσίε, πρέπει να μπορούμε να του εγγυηθούμε και με κάποιο τρόπο ότι θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά του και από οικονομική πλευρά και από πλευρά προσωπικού. Θα το προσέξουμε λοιπόν αυτόν ιδιαίτερα και στη διάρκεια τη συζήτηση και στη διάρκεια τη συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και κρατάμε αυτό που είπε η κυρία Μπερέση. Είναι καλή είδηση ότι φαίνεται να μην απασχολεί εμάς τα μέλη του σε Επιτροπή ΣΕΚΟΝ τόσο πολύ το χρήμα, αλλά άλλα σημαντικότερα ζητήματα. Λοιπόν, για το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ περιορισμένο το χρονοδιάγραμμα. Για το σχέδιο γνωμοδότησης της ΕΚΟΝ 11 Ιουλίου, λίγο μετά θα λήξει προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών και για τη γνωμοδότηση 18 Ιουλίου, εξέταση τροπολογιών και ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ 29 Αυγούστου. Σημειώστε τα αυτά. Και θα ακολουθήσω το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Περιπολογισμών. Να σας ευχαριστήσω όλους ε, όσοι είστε εδώ, να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο μας και επειδή λείπουν οι περισσότεροι για το επόμενο σημείο, διακόπτω για 10 λεπτά τη συνεδρία. Ευχαριστώ.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 So I, I really don't understand. This is such a pity because it seems to be a bit technical. It's so political. I am so important. So the effects is huge importance in the effects as well. I'm amazed that it just got so politicized. I've been since já vím, já jsem říkal, že v pět vyrazí. Když teďka tu ty ryby tady měla být, jako, počkáme, tak on tady není kromě Hybnerova nikdo. Tak.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 Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ε, με το ε, σημείο 14 της ε, ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορά την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή έχουμε ε, λάβει συνολικά 610 τροπολογίες και ε, ήδη ε, το έργο συνεχίζεται προετοιμάζοντας συμβιβαστικές και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή την εισηγήτρια για αυτό το έργο. Παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρατε ήδη κάποια πράγματα και δεν θα ήθελα να το επαναλάβω. Εργαζόμαστε ε, στις, ε, πάνω σε 14 συμβιβαστικές που έχουν προταθεί ε, και από την αρχή, ήδη από την ανάλυση των τροπολογιών, είδαμε ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των ε, μεγάλων πολιτικών ομάδων καθώς επίσης και των συναδέλφων που ανήκουν στην ε, ομάδα διαπραγμάτευσης ε, και μπορώ να πω ότι, έχω, ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του κανονισμού θα έχουμε εν τέλει μια καλή συμφωνία μεταξύ μας. Τα θέματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο αφορούν πρώτον Ε, τα ε, ζητήματα τα οποία ε, σχετίζονται με τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Έχουμε συμφωνήσει να έχουμε το ίδιο σύστημα για την επίβλεψη των CCP της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών εδώ ε, λοιπόν έχουμε μια βασική συμφωνία και έχουμε δημιουργήσει ε, στο πλαίσιο ε, της ΕΣΜΑ μια εσωτερική επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη ε, σχετικά με ε, την ε, νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χθες συμφωνήσαμε σχετικά με την σύσταση της Επιτροπής το μέγεθος αυτής της Επιτροπής Επίβλεψης θα έχουμε μόνιμα και μη μόνιμα μέλη καθώς επίσης μέλη τα οποία θα προσκαλούνται ως παρατηρητές ε, και ε, στο ε, πλαίσιο της η Ρομπέρτα αποφάσισε να συμπεριλάβει πλαίσια όσον αφορά την λογοδοσία της Επιτροπής στην, στο Κοινοβούλιο. Συμφωνήσαμε επίσης πάνω στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα λαμβάνει αποφάσεις ε, μέσω ψηφοφορίας ε, και επίσης πλησιάζουμε σε μια συμφωνία ε, σύνδεση μεταξύ των αποφάσεων και τον ρόλο των επιτηρητών σε αυτή τη νέα δομή της ΕΣΜΑ. Όσον αφορά την επίβλεψη των ε, CCP συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε ε, τα, ε, τα κολέγια και σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την ΕΣΜΑ στο εσωτερικό των κολεγίων και με βάση την αρχή της διάκρισης εργασίας μεταξύ των, της Εθνικής Δικαιοδοσίας και της ΕΣΜΑ έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα αποκαλέψουμε αποκαλέσουμε basketing ε, και ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ε, σύστημα όπου οι εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν την έγκριση της ΕΣΠΑ για ορισμένες αποφάσεις και στη συνέχεια θα υπάρχουν αποφάσεις όπου θα πρέπει να συμβουλεύονται την ΕΣΜΑ και στη συνέχεια θα έχουμε αυτό το καλάθι όπου θα συλλέγονται οι αποφάσεις και ακόμα ε, προβλέπεται και η συζήτηση σχετικά με το ε, σε ποιους ε, τομείς λήψη αποφάσεων θα επισέλθουμε σχετικά με αυτό το καλάθι, Το όσον αφορά τις ε, τρίτες ε, χώρες και την επίβλεψη των κεντρικών συλλαμβανωμένων εκεί. Εκεί θα έχουμε το ίδιο πλαίσιο όπως και με τους αντισυμβαλωμένους τα CCP στην Ευρώπη εδώ έχουμε την ακρόαση, θα ε, είχα το όνειρο στην αρχή να έχουμε την ακρόαση για τους Ευρωπαίους CCP, e ε, κάτι το οποίο δεν έγινε, όμως όσον αφορά τα CCP e των τρίτων χωρών έχουμε ε, το ε, πλαίσιο όπου διακρίνουμε την ομάδα σε T1 που θα είναι λιγότερο συστημικά σημαντικά και για αυτά τα συστήματα ε, η επίκληψη της ΕΣΜΑ, δεν αλλάζει. Στη συνέχεια θα έχουμε το Tier 2 ε, όπου θα έχουμε πιο σημαντικά CCP ε, τα οποία θα υπόκεινται σε απαιτήσει ενισχυμένης επίβλεψης θα πρέπει να επιβάλλεται σε αυτό το θέμα και τρίτον έχουμε την τελευταία κατηγορία που είναι τα ιδιαίτερα συστήματα συστημικά ε, και σε αυτά τα CCP ε, είναι τόσο ισχυρά ε, συστημικά σημαντικά για εμάς ώστε ε, δεν θα τους, δεν θα τους δίνεται αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη τέλος έχουμε κριτήρια τα οποία θα εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ έχουμε την κοινή προσέγγιση, κοινή προσέγγιση και πάνω σε αυτά τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν από την Κομισιόν και από την ΕΣΠΑ όταν θα προβαίνει στην αναγνώριση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση ε, την, ε, το πλαίσιο αυτό και τέλος έχουμε το σύστημα το οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερο το σύστημα μνημονίων συνεννόησης μεταξύ της Ένωσης και των εποπτικών αρχών των τρίτων χωρών όσον αφορά το Tier 2, τα CCP συμφωνούμε στο να αφιερώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα μνημόνια ε, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και όσον αφορά τον σεβασμό αυτών των ε, μνημονίων και επίσης ε, προβλέπουμε και κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχει σεβασμός αυτών των μνημονίων από τις τρίτες χώρες. Επίσης υπάρχει η καθιέρωση ενός κολεγίου επιτήρησης για τις τρίτες χώρες στο οποίο επίσης υπάρχει συμφωνία και τέλος έχουμε ε, επίσης την ανάγκη να υπάρχει μια αξιολόγηση της ε, αναγνώρισης των αποφάσεων. Θα έχουμε ε, κατηγορίες με βάση ε, την ε, ποσότητα οικονομικών εργαλείων που ε, ορίζονται με βάση τα νομίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα συμφωνείται με βάση τα CCP τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά θα αξιολογούνται όσον αφορά την αναγνώριση που θα γίνεται κάθε πέντε χρόνια και επίσης έχουμε ξεκάθαρα κριτήρια για την ε, ΕΣΜΑ, ε, για την κατηγοριοποίηση των ε, CCP, τα οποία ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα. Λάβαμε υπόψη μας στην Επιτροπή Bunch όσον αφορά τον τροπεζικό τομέα και τα πρότυπα που εφαρμόζονται εκεί. Ε, και έχουμε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό πάνω σε αυτά τα κριτήρια. Υπάρχει ακόμα ε, περιθώριο ε, εργασίας όσον αφορά τις κεντρικές τράπεζες έκδοσης των νομισμάτων αυτών για την επίβλεψη των CCP. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ε, διαδικασίας αυτή ε, παραμένουμε NEA ε, όσον αφορά το ζήτημα των κεντρικών τραπεζών και θα γίνουν και κάποιες συζητήσεις σχετικά με το με περαιτέρω κριτήρια τα οποία θα ορίσουμε και εδώ πιστεύω θα βρούμε συμφωνία, θα καταλήξουμε σε συμφωνία και επίσης κάτι το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τη συνάντηση, στη συνάντησή μας με την ΑΦΚΟ θα λάβουμε υπόψη μας την ανάγκη να δούμε αυτή την διάκριση μεταξύ του άρθρου 22 ε, του καταστατικού ε, και της ε, τροπολογίας για την έμειο και ο ρόλος ε, της ε, Κεντρικής Τράπεζας ε, αντικατοπτρίζεται επαρκώς και στις δύο νομικές πράξεις, το οποίο θα το συζητήσουμε στη συνέχεια για να μην σας καθυστερήσω. Ε, ευχαριστούμε πολύ, Ντανούτα. Είμαι σκιώδης εγώ από την πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και όλους τους ε, σκιώδης για την εξαιρετική συνεργασία. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά στην προσπάθεια να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και να αντιμετωπίσουμε πολύπλοκα ζητήματα. και τα περισσότερα από όσα είπατε, Ντανούτα, μας βρίσκουν σύμφωνους. Άρα υπάρχουν ελπίδες ότι θα έχουμε μια καθαρή πλειοψηφία για τα διάφορα ζητήματα τώρα, τα οποία ήδη εσύ ανέφερες, σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, όπως είπες, όλοι επιλέξαμε να παραμείνουμε στις διατάξεις ΕΜΥΡ για να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις με την αθεώρηση της ΕΣΜΑ. Ανεξαρτήτως τώρα των αριθμητικών στοιχείων, η Εποπτική Επιτροπή θα είναι και ένας καλός υποψήφιος στο πλαίσιο αυτών των ε, της αναθεώρησης των εποπτικών αρχών. Σίγουρα σεβόμαστε το γεγονός ότι είναι δύο διακριτή φάκελοι, αλλά θέλουμε να είναι σε πιο ευρύς φορέας, γιατί έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη ιδιοκτησία, και οποίηση αυτού του κοινού καθήκοντος και πιστεύω ότι θεωρείτε και εσείς ότι θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκός αυτός ο φορέας ε, και όχι αντιπροσωπευτικός των εθνικών αφόρων. Για να πω επίσης κάτι θετικό και για την ε, ρήτρα περί ευθύνης και λογοδοσίας. Υπάρχει συνένεση και σε αυτό και στο ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των κεντρικών ε, αντισυμβαλλομένων Πιστεύω θα υπάρχει συνένεση για να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία του ζητήματος και τις διαφορετικές τοποθετήσεις. Αυτή η προσέγγιση, όπως την ανέφερε του μπάσκετινγκ, ίσως να είναι πιο θετική και ενδεδειγμένη για να έχουμε μια ευρεία υποστήριξη. Εγώ πιστεύω επίσης ότι μια ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης πρέπει να συμπεριληφθεί για το μπάσκετινγκ αυτό. Να θεωρηθεί αυτή η λύση προσωρινή που βαθμία θα οδηγήσει σε ένα πληρέστερο σύστημα ευρωπαϊκής εποπτείας. Μίλησε για την κατηγορία κινδύνου και θα αξιολογήσουμε τα άρθρα ακριβώ πώς θα τα κατανείμουμε στα τρία καλάθια η δική μου ομάδα θέλει να μπουν τα περισσότερα στο καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια αλλά λαμβάνουν υπόψη μας και τις διάφορες ανησυχίες για το ρόλο των αρμοδίων αρχών. Να έχουμε δηλαδή μια προσέγγιση δυναμική προς μια ευρωπαϊκή εποπτεία. σε ό,τι αφορά θέμα της Κεντρικής Τράπεζας. Περνάμε ίσως σε μια υβριδική εκδοχή, θα δούμε τι θα γίνει και με μια κατέξοδο της πράξης που μπορεί να διευρύνσω στον κατάλογο. Θέλουμε όμως και έκτα να έχει περιθώρια δράσης σε, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα αυτά άλλωστε σχετίζονται μόνο με την άσκηση των υποχρεώσεων τη έκτη για την πολιτική, ε, συστήματα πληρώμα κτλ. Ε, δεν είναι και εύκολο να το πλαισιώσουμε το σύστημα. Έχω καταθέσει τροπολογίες. Θα τις επεξεργαστούμε. Και το θέμα αυτό σχετίζεται και με το επόμενο σημείο της Μερσιδέας με το άρθρο 22 για την αναγνώριση των χωρών. Νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλειά, πλησιώντα καλύτερα το τύριν και διατηρώντας και την θέση της Κομισιόν για ένα ειδικό καθεστώς για να δούμε τι θα γίνει με την, με την κατάσταση το σύστημα νομίζω ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Δεν είναι μόνο στο χαρτί μια επιλογή. We are a, νομίζω ότι συγκλίνουμε προς μια λογική ε, λύση, προς ένα λογικό συμβιβασμό, προσθέτοντας και κάποιες διευκρινήσεις που ελπίζω να ε, περάσουν οι σχετικές στις αιτηλογικές σκέψεις. Γι' αυτό το νέο σύστημα steering με ειδικά χαρακτηριστικά για κάποια γερικά παράγωγα για να μειωθούν οι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά τα συστήματα συμψηφισμού και υπάρχει εφαρμοστική βάση απόφασης οδυναμίας ε, που έχει εγκρίνει η Κομισιόν ήδη. Απλά με τη σκέψη θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο για να διαταράξουμε και να προκαλέσουμε αχρία στο κατακαιρματισμό της αγοράς. Τέλος, ό,τι αφορά την αναθεώρηση, καταθέσαμε τροπολογίες για μια ε, μεγαλύτερη αναλογικότητα για τα αναγνώριση τρίτης χώρας, δύο χρόνια, λέμε ότι για κάποιε περιπτώσεις πρέπει να ισχύει ένα όριο και για άλλες πέντε χρόνια. Αυτές είναι οι τροπολογίες ουσιαστικά που έχουμε καταθέσει. Είναι καλό το κοινοκείμενο, είναι μια καλή βάση, πιστεύω. Θέλω να ευχαριστήσω την Τανούτα και όλους τους άλλους συναδέλφους. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία μέχρι τώρα. Εσείς ποιον εσείς θα εκπροσωπήσετε την ΚΕΙ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Μιλάω εξ ονόματος της Κέι Σουίμπερν, η οποία ζητά συγγνώμη διότι δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα και θα σας διαβάσω τη δήλωση εκ μέρους της. Καταρχάς ευχαριστεί την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους σκιώδεις για τα σχόλια που έχουν κάνει μέχρι τώρα οι τροπολογίες ε, που υπέβαλαν ε, οι σκιώδεις του ECR και οι συνάδελφοι αντανακλούν κάποιες βασικές θέσεις του ECR. Το ρόλο του εθνικού επόπτη, τη σημασία ε, του σεβασμού των ε, κρατών μελών εκτός Ευρωζώνης και να υπάρχει και ένα αποδοτικό σύστημα. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες υπευλήθησαν από συναδέλφους που θεωρούμε ότι υποστηρίζουν αυτές τις θέσεις, τροπολογίες από όλο το Κοινοβούλιο που επισημαίνουν πόσο σημαντική είναι η συνεργασία ε, εποπτική συνεργασία και την γιατρή, η CCP τρίτων χωρών και η πρόταση του κυρίου Γκαλτιέρη για να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με CCP τρίτων χωρών. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμε προτάσει για ένα θέμα το οποίο έχει γίνει ιδιαίτερος πολιτικό. Όσον αφορά την Εποπτική Επιτροπή, υποστηρίζουμε τι τροπολογίε του κυρίου Γκαλτιέρη για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία του συγκεκριμένου φορέα και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν και δύο περαιτέρω αντιπρόεδροι από πλευρά Άλντε θα το εξετάσουμε. Ε, όσον αφορά το θέμα του ρόλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως ήταν ιδιαίτερο για, την, ε, ε το ECR, κυρίως για τη δυνατότητα που δίνεται στην ΕΚΤ να επιβάλλει βέτο σε κάποιες αποφάσεις. Ε, μας ενδιαφέρει ο ρόλος του CBI που έχει κυρίως στόχο την άσκηση της νομισματικής πολιτικής την ανάγκη ε, για μια ε, διαδικασία συμμόρφωσης την υποστηρίζουμε ε, κυρίως για κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωζώνης και την εισαγωγή ε, CCPs όπου ε, αυτό μας αφορά. Μας ανησυχεί η τροπολογία 61 που εισάγει την ιδέα της δράσης της CBI μόνο σε εξαιρετικές συνθήκες. Αλλά υποστηρίζουμε την συζήτηση που θα γίνει στις σκιώδεις συγητές για να βρούμε μια λύση. Τώρα, την πολιτική όσον αφορά την ε, ε, έδρα. Δεν θεωρούμε ότι είναι ε, υπεύθυνη αυτή η επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα προτείνει κατακαιρματισμό, θα οδηγήσει μάλλον σε κατακαιρματισμό και θα έχουμε ένα λιγότερο εύρο στο σύστημα CCP που δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστική. Υποστηρίζουμε λοιπόν την τροπολογία 476 του κυρίου Λούτβιχσον σε αυτή την περίπτωση. Αναγνωρίζουμε τις τροπολογίες οι οποίες έχουν μια λογική και ένα πλαίσιο, ιδιαίτερα την 477 του Άλτε, την 478 της Νίνα Γκίλ και την 479 του Τόμας Μαν. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε το περιεχόμενο των τροπολογιών που τονίζουν ε, ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικός ε, ε, μετριασμός του κινδύνου σε αυτή την περίπτωση και ότι θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση αντικτύπου πριν ληφθούν περαιτέρω βήματα. Το ECR δεν υποστηρίζει την άποψη του κυρίου Κλίντ στην 474 ότι το CCP ε, ε, κατηγορίας 2 δεν θα πρέπει να βρίσκεται διότι εδώ, διότι θα μειώσει οποιαδήποτε η αναλογικότητα στο εποπτικό σύστημα και αποτελεί κίνδυνο για το πορό σύστημα. Η συνάδελφο χαίρεται που προχωρούν καλά οι συνεδριάσει των σκιωδών, προσβλέπει σε συνεργασία πριν από την ε, ε, ψηφοφορία με τους σκιώδες και τις περαιτέρω τεχνικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάτσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, την εισηγήτρια και τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Ήταν πολύ αποτελεσματική και φυσικά αυτό ισχύει και για τους κοιότης. Καταρχάς, για κάποιες βασικές προτεραιότητες για μας. Όσον αφορά την εσωτερική εποπτεία των CCP, συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να περάσουμε προς ε, μία αναγνώριση ενός συστήματος εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κοινωνικών Αξιών και Αγορών. Γι' αυτό ακριβώ και υποβάλαμε τροπολογίες για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η δομή αυτή στην πράξη. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα ε, μέλη της Εποπτικής Επιτροπής από όσα αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης και γι' αυτό ακριβώ έχουμε προτείνει δύο αντιπροέδρους επιπλέον. Θα υποστηρίξουμε ένα πρόεδρο και ε, συγκεκριμένα μόνιμα μέλη της Επιτροπής. Επίσης θέλουμε να έχουμε συνέπεια του κειμένου με ε, την συμφωνημένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάκτηση ποσών και την εξυγίανση των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών. Επίσης θεωρούμε ότι οι κίνδυνοι που λαμβάνονται ε, υπόψη από τις αρχές τρίτων χωρών για το κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση των κεντρικών αντισυμβαλόμενων σε αυτόν τον κανονισμό, συγκεκριμένων των ε, χρηματοπιστωτικών, επιχειρησιακών και, κυβερνο... Ε, και κινδύνων στο κυβερνοχώρο. Επίσης θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται με τους κεντρικούς ε, αντισυμβαλόμενους, να γίνονται έλεγχοι τακτικά ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ετοιμότητα σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Όσον αφορά για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους τρίτων χωρών, οι περισσότερες ομάδες συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την ε, ανάκληση της αναγνώρισης κάποιων κεντρικών αντισυμβαλόμενων που παρουσιάζουν ε, συνεχή συστημικό κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη Ένωση. Στι τροπολογίε μα θέλουμε να διευκρινίσουμε τη διαδικασία εφαρμογή αυτού του μηχανισμού, τονίζοντα ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν μεταξύ μια απόφαση ανάκληση και τη εφαρμογή τη. Αυτό θα πρέπει να προσφέρει στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει τον απαραίτητο χρόνο για να επαναδιαπραγματευτούν συμβάσει, να προσπαθήσουν να μετριάσουν τυχόν επιπλέον κινδύνου που θα προκύψουν από τον κίνδυνο αυτό και ε, τη δυνατότητα εγκατάστασης ε, της επιχείρησης εκαθάρισης. Κάποιες υπηρεσίες ε, στις διαδικασίες κεντρικού αντισυμβαλόμενου που έχουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει να ε, ανακαλούνται οι αδειές τους, η αναγνώρισή τους. Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση κάθε κεντρικού αντισυμβαλόμενου ε, για να μπορέσουν να διασφαλίσουν σε ποια κατηγορία θα εμπίπτει. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες ε, οι οποίες θα μοιράζονται μεταξύ κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2 και αυτό θα δίνει στις επιπτικές αρχές και καλύτερο έλεγχο για τις διάφορες υπηρεσίες και θα υπόκειται και σε περαιτέρω απαιτήσει. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο ακολουθεί τη σωστή προσέγγιση και ε, υποστηρίζω το επικοδομητικό έργο που έχει γίνει μέχρι τούδε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια Ντανούτα, συμφωνούμε πολύ με την αξιολόγησή σου ότι θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω εποπτεία και ε, επιτήρηση γιατί υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι για αυτούς τους οργανισμούς. Επίσης, συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση όπου η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα μπορεί να εφεσιβάλλει αποφάσεις ε, των ε, αρχών των κρατών μελών. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω τροπολογίες στο άρθρο 21A3 ε, το οποίο επιτρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες εποπτικές δράσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και να εφαρμόζονται αυτές οι δράσεις σε περίπτωση αδράνειας από τους εθνικούς, ε, τις εθνικές αρχές ή την τροπολογία στο 21A6 που ενισχύει το ρόλο της ΕΣΜΑ σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ εθνικών αρχών. Κάτι άλλο στο οποίο συμφωνούμε μαζί σου είναι ότι η ενασχημένη εποπτική διαδικασία των κεντρικών τραπεζών θα πρέπει να τη χάνει και τη ανάλογη ισορροπία. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε διαβούλευση τη κεντρική τράπεζα ε, πριν εφαρμοστούν μέτρα όσον αφορούν τη ρευστότητα τι εγγυήσει και τι κεντρικέ απευθύνσει των οργανώσεων αυτών σε σχέση με τα όσα έχουμε στο σχέδιο κειμένου σου και στην πρόταση τη Επιτροπής. Εδώ διαφωνούμε λίγο. Τα πιθανά προβλήματα ρευστότητα μπορεί να επηρεάσουν τα συστήματα πληρωμών σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικέ αναταραχέ, αλλά δεν προβλέπουμε ότι οι κεντρικέ αρχέ θα πρέπει να ζητήσουν από ένα κεντρικό αντισυμβαλόμενο να ζητήσει νέα άδεια τράπεζα. Αυτό φυσικά θα πρέπει να το δούμε βάσει και των στόχων των, ε, της παρακολούθησης των στόχων πολιτικής. Αυτό που με ανησυχεί πάντα είναι ότι όταν προσπαθούμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και περισσότερες αρμοδιότητες στις κεντρικές τράπεζες μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Επίση, συμφωνούμε ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει μία από τι αδυναμίε του παρόντο πλαισίου, διότι το καθεστώ βασίζεται ε, στι εποπτικέ αρχέ των τρίτων χωρών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θεωρούμε ότι οι γενικέ γραμμέ είναι κατάλληλο και αναλογικό το σύστημα, αλλά συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι το κείμενο του επίπεδου ένου θα πρέπει να δει λίγο καλύτερα τα κριτήρια βάσει των οποίων ε, γίνεται ταξινόμηση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων σε τρει κατηγορίε. Εδώ τροποποιούμε και το άρθρο 21.2c για να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράξη κατεξουσιοδότηση για να καθορίσει αυτά τα κριτήρια και ενισχύουμε και τις ε, εξουσίες της ΕΣΜΑ για να μπορεί να επιβάλλει και ρυθμιστικές απαιτήσεις σε ε, πιθανά συστημικά προβλήματα με συμβελόμενους τρίτων χωρών ε, σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τις κεντρικές τράπεζες. Και κάποιες άλλες προτάσεις για τα νέα CCP. Προτείνουμε μια τροπολογία στο 25.2 ββ που θα μπορεί να επιβάλλει νέα θηγατρική για να πάρει άδεια τράπεζα σε τρίτε χώρε. Όσον αφορά τη δομή τη Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καταλαβαίνουμε την προσέγγισή σου, αλλά ανησυχούμε λίγο ότι μπορεί να δημιουργήσουμε πολύ ε, μεγάλη γραφειοκρατία και επομένω προτείνουμε κάτι εναλλακτικό όπω γνωρίζει, Ξέρουμε ότι υπάρχει η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, αλλά ε, πιστεύουμε ότι πριν από την έγκριση τη αναθεώρηση. ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής μπορεί να γίνουν από τον πρόεδρο και τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΣΜΑ. Ε, βλέπω ότι είναι και ο μάλλον ο κύριος Λουκ έφυγε, ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε. Αντιλαμβάνομαι όλες αυτές τις ερωτήσεις για τον κατακαιρματισμό της αγοράς, αλλά θα ήθελα να πω κυρίω στο ECR ότι οι δημοκρατίε μας είναι καταχειρηματισμένες. Δεν έχουμε μια παγκόσμια δημοκρατία και επειδή θέλουμε οι αγορές να υποβάλλονται στη δημοκρατία και όχι το αντίστροφο, είναι λογικό ότι εφόσον δεν υπάρχει μια παγκόσμια δημοκρατία, δεν υπάρχουν και παγκόσμιες αγορές. Υπάρχει κατακαιρματισμό δεδομένου ότι υπάρχει κατακαιρματισμένη δημοκρατία, αλλά προέχει η δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάθη δεν είναι εδώ. Από το EFTD δεν θέλει να μιλήσει κανείς. Κύριε Άνεμανς, θα μιλήσετε. Κυρία Βίνη, ξέρετε το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Ο συνάδελφος Βόλφ Κλίντς μου ζήτησε να διαβάσω κάτι. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο συνάδελφο Βολκ δεν μπόρεσε να έρθει στην συνεδρία σήμερα το απόγευμα και μου ζήτησε να σα διαβάσω την εξή εξήγηση για να υποστηρίξει την ε, τροπολογία του 474, στην οποία ζητάμε κατάσταση ε, των αντίστοιχων ε, ε οίκων εκαθάρισης ζητά ε, δεδομένης απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε μεγάλο αντίκτυπο των ευρωπαϊκών συστημάτων στη δυνατότητα να διεξάγουν τα καθήκοντά του ω κεντρική τράπεζα για το ευρώ και επιπλέον ότι θα υπάρχουν πολύ σημαντικέ τρευλώσει ε, για τους ε, Κεντρικού αντισυμβαλόμενου του Ηνωμένου Βασιλείου και μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη αύξηση ρευστότητα ε, στον ε, χώρο τη Ευρωζώνη. Ε, τα όσα προτείνει η συγγήτρια αποδυναμώνουν αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να έχουμε συστημική σημασία για τι περιφερειακέ εργασίε των CCP και να έχουν αντίκτυπο αντί για τη συστημική σημασία του CCP για το ευρώ συνολικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει πλέον να δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και επομένω η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εξαρτά την χρηματοπιστωτική της σταθερότητα από την καλή βούληση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητά της να προστατεύσει τη σταθερότητα του νομίσματός του. Brexit σημαίνει Brexit. Οι οίκοι καθάριση που έχουν συστημική σημασία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμεύονται από το κοινοτικό κεκτημένο και επομένω θα πρέπει να μετεγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τουλάχιστον στον ΕΟΧ σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να συμμετέχει στον ΕΟΧ, ε, δεν θα πρέπει να αλλάξει τίποτα. Αυτό θα μπορούσε επίσης να αποτελήσει και πολύ καλό ε, αντίβαρο στις ε, διαπραγματεύσεις για τον Brexit για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά για τον δυνητικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις, υπάρχουν επιπλέον τροπολογίες του κυρίου Γκλίνκ, Κλίντς, ώστε μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2021 που ίσως να έχουμε τον Brexit να υπάρχει εκαθάριση των νέων επιχειρήσεων εντός ε, του ΕΟΧΟ όλα τα οικονομικά συστήματα. Ακόμα και αν χάσουν 10 χρόνια ή αργότερα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά το, το Brexit και δεν θα πρέπει να γίνει εκ νέου καθάριση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητά το λόγο. Υπερβάσπερες. Ευχαριστώ. Κυρία Συγήτρια, σας ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο πραγματικά Θέλησατε να δώσετε το ρυθμό σας και νομίζω ότι το περιεχόμενο της συζήτησης σας βοηθά να προχωρήσετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν εξέτασα με πάσα λεπτομέρεια τις συμβαστικές προτάσεις ακόμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ως προς την ουσία περιλαμβάνονται τα πάντα. Έχουν και κάποιες ανησυχίες, οι οποίες θα υπενθυμίσω και κυρίως ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι δεν συζητήσαμε. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις εξουσίες της ΕΣΜΑ. Συμφωνούμε μαζί σας ότι θα πρέπει να ε, δούμε το υποπτίας ε, το κεντρικό της συμβαλόμενο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το είδαμε στην εξέταση του κειμένου σας και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν αναφέρεται νομίζω το θέμα των ειδικών εξουσιών σε περίπτωση κατεπήγοντος. Διότι έχω την εντύπωση ότι αν υπάρχει συστημικός κίνδυνος θα πρέπει να μπορούμε να προβλέψουμε και κατεπήγουσες περιπτώσεις ώστε να μπορεί να παρέμβει έσμα ε, υπό συγκεκριμένε συνθήκες. Και όσον αφορά το θέμα της δημοκρατίας ε, δεν μπορώ να αντισταθώ, πρέπει να απαντήσω. Όταν έχουμε παράγοντες της αγοράς ε, που δεν γνωρίζουν κανένα κατακαιρματισμό και δημοκρατίες οι οποίες εξακολουθούν να είναι κατακαιρματισμένες ε, στο όνομα της εθνικής εξουσίας ε, Πολλά μπορεί να είναι κοινά, μπορεί να, πολλά να μεταβιβαστούν και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό που έχει το ρόλο να το διορθώσει αυτό το θέμα. Να υπάρχει μια ευρωπαϊκή εποπτεία και νομίζω ότι η παρέμβαση του Κοινοβουλίου είναι πλήρω υπεύθυνη λύση σε αυτή την περίπτωση. Κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο έχει σχέση και με την αναθεώρηση των ε, Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Συμφωνώ με αυτό που προτείνεται. Καταλαβαίνω ότι αυτό που προτείνεται είναι μια συγκεκριμένη ε, αρχή για την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλόμενων. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να δούμε μαζί με την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και κυρίως τα όσα θα δούμε στην αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και θα δούμε και το θέμα της διακυβέρνησης και ίσως εδώ ένας εκ των ε, αντιπροέδρων του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος αυτού του Συμβουλίου το οποίο συστήνεται για την εποπτεία. Όσον αφορά τον ιδανικό αριθμό των μελών ε, σε αυτό το όργανο, δεν έχω άποψη. Ξέρω όμως ότι ένα εκτελεστικό όργανο για να είναι αποτελεσματικό δεν θα πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μελών και υπάρχει μια κλίμακα αξιών για τα όσα έχουμε όσον αφορά τη λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας ή άλλων ε, αντίστοιχων οργανισμών. Δηλαδή, αυτό που λειτουργεί καλά το γνωρίζουμε και αυτό που δεν λειτουργεί πολύ καλά επίση το γνωρίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι από αυτά που λειτουργούν καλά. Αποτελείται από έξι μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν συγκεκριμένε αρμοδιότητε. Δεν ξέρω ποιο είναι ο ιδανικό αριθμό, δεν έχω εικόνα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Ε, επιτρέποντας βεβαίως να υπάρχει και ε, συνδυασμός με τη νέα διακυβέρνηση που θα έχουμε στην ΕΣΜΑ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Τζένιφερ Ρόμπερτσον, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω την πολύ καλή δουλειά του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Έχει σημειωθεί πρόοδος. Χαίρομαι που βλέπω τη στήριξη στο Κοινοβούλιο όλες τις βασικές αρχές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά ε, τις διατάξεις για την αγνώριση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων τρίτων χωρών ε, είναι καλό να υπάρχει αυτή η προσέγγιση του tiering των βαθμίδων. Επίσης καλό είναι που υπάρχει ανεξάρτητη εποπτική αρχή με την σωστή στελέχωση υπό, στο εκπρόσωπο της ΕΣΜΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών και Αγορών. Υπάρχουν τώρα κάποιοι άλλοι τομείς, αν καταλάβαμε σωστά βέβαια το σχέδιο της έκθεσης, όπου θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να ξανασκεφτεί κάποια πράγματα και ίσως να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη συγκρίσιμη συμμόρφωση. Συγκρίσιμη συμμόρφωση, τι σημαίνει, πώς ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος μιας τρίτης χώρας ε, ε, εκπληρεί το σχέδιο όχι μιας τρίτης χώρας, ε, αλλά το πλαίσιο της Ένωσης. Ε, και αυτό πρέπει να λέγεται ξεκάθαρα για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μήπως έμεσα εισαγάγουμε διπλή εποπτεία για κεντρικό αντισυμβαλό. Θα πρέπει να βλέπουμε αν είναι η συστημική σημασία του αντισυμβαλόμενου μεγάλη και αν συμμορφούνται προς όρους 2β και το και Αν δεν αρκεί αυτό, θα πρέπει και άλλοι όροι να πρέπει να πληρούνται για να μην τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών, θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα το δικαίωμα των κεντρικών τραπεζών και ο ρόλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλόμενων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρόμαστε που προβλέπεται ένας κεντρικός ρόλος για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ίσως όμως έχουμε αυτή τη, το σύστημα βαθμίδων και για τους αντισυμβαλλόμενους από τις χώρες μέλης Ένωσης. Αυτό μας ανησυχεί. Δεν ξέρω αν κατάλαβα και καλά την κυρία Χούμπνερ, αλλά νομίζω ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια μετακίνηση ως προς αυτό συστημικά σημαντική είναι όλοι οι κεντρικοί συμβαλόμενοι της Ένωσης για την Ένωση. Άρα όλοι θα πρέπει να υπάγονται στην εποπτεία από την ΕΣΜΑ χωρίς διαφοροποίηση με βάση το προφίλ κινδύνου. Thank you. Yeah, you correct. Ευχαριστώ. Ναι, γι' αυτή ακριβώ είπαμε ότι θα ακολουθήσουμε την προσέγγιση του μπάσκετ. Κυρία Χούμπνερ. Προς τον κύριο Βόλφ Κλίντς να πω. Προετοιμάζεται ένας κανονισμός που θα διαμορφώσει τις αγορές μέσω και μακροπρόθεσμα. Όχι ένας κανονισμός που θα αντιδράσει ad hoc συμβάντα. Αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι η πρόθεση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό και ανταποκρινόμαστε στο αίτημα των διαπραγματευτών του Brexit. Είναι σημαντικό να μην προεξοφλήσουμε στον κανονισμό το δυνητικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά την αποχώρηση της και το τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν προεξοφλούμε και δεν προτείνουμε ad hoc μέτρα που θα μπορούσαν να λαμβάνονται σε αναδυόμενες καταστάσεις. Μην παρανοήσουμε το ρόλο του κανονισμού και του κοινοβουλίου και του έργου μας πάνω στον κανονισμό αυτό. Επίσης, αυτό το σύστημα βαθμίδων, το tiering, στην πρώτη εκδοχή πριν τα Χριστούγεννα, που προσπαθούσα έτσι να συμμετρήσω ε, την άποψη των υπολείπων και ήταν αρνητική και δεν συνέχισα βέβαια. Κάποιος με έπαιρνε και από τηλέφωνο που έλεγε ότι μάλλον θα ήταν καμιά καλή προσέγγιση αλλά μπορείτε να κοιμάστε ήσυχη Επιτροπή. Δεν θα ισχύσει. Εκτός εάν το προτείνει το Συμβούλιο. Αν έχει καλά επιχειρήματα θα το ξαναεξετάσουμε, αλλά δεν μας φαίνεται πιθανό κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση. Μάλλον παρανόηση έγινε. Θα δω τη διατύπωση, αλλά δεν βλέπω να έχει κάποιος άλλος αμφιβολίες για αυτή τη διπλή αποπτία. Φαντάζομαι μιλάτε για κάποιε τροπολογίε. Υπάρχουν πολλέ τροπολογίε που δεν θα καταλήξουν σε συμβαστικέ. Μπορεί να είναι μια τροπολογία μεμονωμένη, αλλά καλό θα μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το ποια συγκεκριμένη η τροπολογία είναι αυτή. Σε τέφα το μέγεθος. Μέγεθος των επιτροπών Αυτά είναι αντικείμενα μελλοντική διαπραγμάτευση κατά με. Χθε αποφασίσαν μπορεί να μην με κάτι άλλο να είναι. Έπρεπε να συμφωνήσουμε σε ένα νούμερο. Απλά ε, κάποια πρόταση κάναμε που θεωρούμε ότι είναι λογική. Το ξέχασε ο Ρομπέρτο. Αλλά έλεγε ο Ρομπέρτο να είναι μια γυναίκα, να είναι κάποιο εκπρόσωπο μια μεγάλη χώρα, κάποιο εκπρόσωπο μια μικρή χώρα κτλ. Να υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στο σώμα αυτό. Θα δούμε. Ελπίζω να μην υπάρξουν πολιτικέ διαφωνίε από αυτού. Συμφωνήσαμε επίση ότι θα πρέπει να δούμε το μέγεθο. Κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν πολύ μεγάλο. Αλλά είναι προσωρινό το μπάσκετινγκ αυτό. Εμείς θέλουμε ευρωπαϊκή εποπτεία στο τέλος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μια νυχτή. Πρέπει να υπάρξει ένα σταδιακό σύστημα, phasing in, σταδιακής υιοθέτησης της ευρωπαϊκής εποπτείας. Η ΕΣΜΑ ίσως να μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες της διαδικασίας, αλλά σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση γιατί είναι πρώτη φορά που ασχολείται, είναι αρχάρι αν θέλετε, ε, προς αυτό το τομέα. Άρα το μέγεθος θα εξακολουθήσει να συζητείτε. Σε ό,τι αφορά την ΕΣΜΑ συγκεκριμένα και όχι την Κεντρική Τράπεζα, για την ΕΣΜΑ τα μνημόνια, τα λίγη πληροφοριών είναι σημαντικό. Εκεί εστιάζουμε, αλλά τα μνημόνια είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια τη ΕΣΜΑ, τη Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. τοπική Κομισιόν. Όταν ο επόπτη δεν φέρνει αποτελέσματα από την άλλη πλευρά, δεν αντιδρά σε καταστάσεις ε, που αναδύονται, για παράδειγμα, τότε υπάρχει και το δεχόμενο να ανακληθεί η αναγνώριση του κεντρικού αντισυμβαλωμένου. Προβλέπουμε τέτοιες, τέτοιες δυνατότητες σε περίπτωση δυσκολίας. Επίσης θέλω να πω ένα ευχαριστώ, το έκανε και ο Ρομπέρτο, το λέω και εγώ, ένα ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους, αλλά και τους ε, βοηθούς μας, τους συνεργάτες μας, τους ε, συμβούλου μα βοηθούν σε τεχνικό επίπεδο. Πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερο στη βοήθειά του. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα. Και πριν φύγουμε, να έχουμε ολοκληρώσει. με την νομοθεσία αυτή για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και για αυτό το χαρτοφυλάκιο, για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών υποπτικών αρχών δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να προεξοφλήσουμε τις ιδέες και τις απόψεις. Έξω και αυτή η διάρθρωση που είναι εσωτερική διάρθρωση. Και σε πολλές άλλες ε, περιπτώσεις ε, ε, προσπαθούμε να αποφύγουμε, να προδικάσουμε τα πράγματα. Αλλά το σημειώνω αυτό που είπατε is well I, talked about uh, ESMA you mean no no emergency emergency ε, μίλησα για την ΕΣΠΑ ε, όχι όσον αφορά το ECBI σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης είναι πολύ καλά αλλά εγώ κατάλαβα ότι ε, μιλούσατε για την ΕΣΜΑ Θα το συμπεριλάβουμε και αυτό, θα εργαστούμε πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται να υπάρξουν τα πάντα. Χθες, ε, το, ε, προχθές μάλλον, ε, το συζητήσαμε αυτό και κάνουμε μία διάκριση μεταξύ του άρθρου 22, 22 και το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο ούτως ώστε να συμπεριλάβουμε τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να παρέμβει έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών ε, διότι ε, δεν γίνεται να το έχουμε αυτό ε, στο κανονισμό ΕΜΗΡ και όσον αφορά το άρθρο 22 θα ήταν ο καλύτερος τρόπος, τρόπος για την Κεντρική Τράπεζα να περιορίσει και να αντιδράσει σε περίπτωση που υπάρχουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Αυτή είναι η βασική ανησυχία. Ευχαριστώ ε, πολύ. Υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίες, ε, όπως ε, για παράδειγμα τη δυνατότητα αντίδρασης της κεντρικής τράπεζας σε περίπτωση εκτάκτης ανάγκης, όμως το βασικό εργαλείο για αυτό είναι το καταστατικό. Ακόμα συζητάμε πάνω σε αυτό. Χθε είχαμε την πρόταση και τώρα θέλουμε να έχουμε καλύτερη έκφραση στο κείμενο πάνω σε αυτό. Δεν πήραμε κάποια απόφαση χθες. Έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες. Είναι μια εναλλακτική την οποία ε, σκεφτόμαστε. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μια τέτοια ε, τροπολογία. Δεν είναι μυστικό. Οπότε το θέμα είναι ποια θα είναι η τελική πρόταση της συμβιβαστικής. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. και συγχαρητήρια στο προσωπικό για την υποστήριξη. Έχουμε ένα ε, γεμάτο ε, ε, ε διάγραμμα. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 16 ε, Μαΐου του 2018. Θα πρέπει να γίνει μια επιβεβαίωση αυτού όμως ε, η ομάδα έχει εργάζεται σκληρά πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι θα ε, τα καταφέρουμε. Αν ε, δεν είμαστε έτοιμοι ως τότε, τότε θα το αναβάλουμε για λίγο, αλλά το αν θα γίνει στις 16 Μαΐου ή μια-δυο εβδομάδες αργότερα Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε εν καιρό την ανάγνωση, ούτω ώστε να αρχίσει ε, στο πλαίσιο αυτής της προεδρίου, προεδρίας ε, ο τριμερής ε, διάλογος. κρατούμε λοιπόν την ημερομηνία ψηφοφορίας που έχουμε για την ώρα, διότι μας δίνει το κίνητρο να επιταχύνουμε και στη συνέχεια ε, εγκαίρως θα επιβεβαιώσουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε λίγο νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε, οπότε η, η επόμενη συνάντηση είναι κοινή συνάντηση με την Επιτροπή ΕΦΚΟ, οπότε θα περιμένουμε. Έχουμε 15 ε, λεπτά διάλειμμα